Prendiamo posto. Ξεκινάμε. Prendiamo posto. Olenicka is the only socialist today. the strong socialist representation. Ιδιαίτερα ισχυρή σοσιαλιστική παρουσία. Bene. Se siamo d'accordo diamo inizio alla commissione, do il benvenuto a tutti. Λοιπόν, ξεκινάμε, σας καλωσορίζω όλους. Για τεχνικούς λόγους να σας ενημερώσω ότι λείπουν σήμερα τα φιλανδικά και τα σλοβενικά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. να συγχαρώ την Ιταλική ομάδα του Ράγκμπι για τη μεγάλη τους νίκη το Σάββατο. Ελπίζω ότι έχετε συνέλθει από τις μεγάλες γιορτές και θα μπορέσετε να διευθύνετε τις εργασίες μας με επαρκώς. Ευχαριστώ Άγνιο. Λοιπόν, έλεγα και ζητώ συγγνώμη ότι σήμερα δεν έχουμε μαζί μας διευμηνία προς τα φιλανδικά και τα σλοβενικά. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις λοιπόν. Δεκτή η ημερήσια διάταξη. Θυμίζω επίσης ότι μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις, θα γίνουν δεκτά και τα πρακτικά της 7ης Φεβρουαρίου. Ε, θυμίζω επίσης ότι ε, θα αναμεταδοθεί στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συγγραφείς της μελέτης για τα μέτρα της αγοράς στη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική. Ποια πρέπει να είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Ιζαμπέλ Μπαρντάζη, τον Αλμπέρτο Γκαρίδο και οι δύο ερευνητές ε, του, του Πανεπιστημίου, του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Μαδρίτης. Τους δίνω αμέσως το λόγο, τους υπενθυμίζω ότι έχουν 20 ε, λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν την παρουσίασή τους. Καλωσορίζω επίσης και τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Μπαρντάζη και Γκαρίντο έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια, είναι ομαδική προσπάθεια συμβούλων από τη Μαδρίτη. Έχουμε συμβούλους από πολλές χώρες. Θα χρησιμοποιούσα στο πρώτο τμήμα της παρουσίασης την αγγλική γλώσσα και θα συνεχίσει η συνάδελφός μου στα ισπανικά. Τα εξή είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, τα παρουσιάζω συνοπτικά. Πρώτον, θα ήθελα να μιλήσω για το πλαίσιο, την αύξηση της κινητικότητας στον τομέα των τιμών, τη μακροπρόθεσμη τάση ή την αυξητική, την πειθαρχία στον ΠΟΕ, την έκθεση στη διεθνή αγορά, στην παγκόσμια αγορά, τη σύνδεση με τη βιοενέργεια, την πολιτική για τη βιοενέργεια, ε, την ε, υπερσυγκέντρωση του λιανικού τομέα και του βιομηχανικού τομέα και την δυνατότητα χρήσης ε, των ηλεκτρονικών μέσων στην μελλοντική ΚΑΠ. Τρεις είναι οι παράμετροι για αυτή την προσπάθεια. Καταρχάς οι τιμές είναι θα έλεγα στοιχεία πληροφόρησης Δεύτερον, οι παραγωγοί θα πρέπει να στραφούν καλύτερα στις αγορές και να μάθουν να διαχειρίζονται καλύτερα τις αγορές και τους κινδύνους. Ε, τρίτον, ε, τα μέσα διαχείρισης της ιδιωτικής αγοράς ε, δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αρκετά στο παρελθόν, ενώ θα πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει στο μέλλον. βλέπουμε κάποια παραδείγματα και κάποιες καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων μπορούμε να μάθουμε πόσο χαμηλά θα πέσουν οι τιμές. Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο πολιτικής θα πρέπει να λειτουργήσουν προληπτικά και όταν έχουμε πολύ χαμηλές τιμές θα πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε τέτοιες αποφάσεις μέσα σε ένα πλαίσιο θα έλεγα αβεβαιότητας. Θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής εδώ προτάσεις. Καταρχά, έχουμε σαν θεμέλιο τα διαρθρωτικά μέτρα της αγοράς και πρόσβαση στα τρόφιμα. Πρέπει να υπογραμμίζουμε εδώ ότι οι τομείς της αγοράς καταρχάς στον τομέα της τιμολόγησης λειτουργούν θεωρητικά τουλάχιστον με κανονικό τρόπο αλλά δημιουργούνται και άτακτες εισαγωγικά περιπτώσεις. Χρειάζεται λοιπόν σωστή ενημέρωση για την κανονική κατάσταση στην αγορά. Χρειαζόμαστε προληπτικά μέτρα για να προπαρασκευάσουμε τον συγκεκριμένο τομέα να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις. Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίδρασης. Αυτή είναι η στάση που θα πρέπει να κρατήσουμε. Βλέποντας τώρα τα διαρθρωτικά μέτρα και την πρόσβαση στα τρόφιμα, χρειαζόμαστε μια καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Καλύτερες επαφές και συμφωνίες, καλύτερος με τους παραγωγούς, με τις οργανώσεις των παραγωγών, με τις αντιπροσωπείες των παραγωγών, χρήση των πλεονασμάτων όταν αυτά υπάρχουν μέσω βοήθειας προς ε, πληθυσμούς με, με προβλήματα δυνητικά κτλ. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα προληπτικά μέτρα. Εδώ έχουμε τα μέσα διαχείρισης των κινδύνων των αγορών των γεωργικών προϊόντων. Κάλυψη λοιπόν των αγορών, των αναγκών των αγορών, ασφαλίσεις και κάποια νέα μέσα Εν πάση περιπτώσει αυτά τα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν το εισόδημα μπορούν να συνδυαστούν με συγκεκριμένες πληρωμές ή και με μέσα διαχείρισης των αγορών σχετικά με την αποθήκευση των προϊόντων και την πρόθεση των προϊόντων. Τα μέτρα λοιπόν που προτείνουμε για την ΚΑΠ στο μέλλον είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να είναι σχετικά ταυτόσιμα θα έλεγα ανεξαρτήτως της συγκυρίας. Καταρχάς, στόχοι μας θα πρέπει να είναι η λειτουργία της σωστότερης αγο... λειτουργίας της αγοράς μάλλον. Η μηχανή... Οι μηχανισμοί τους οποίους έχουμε στην διάθεσή μας θα πρέπει να λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς εξαιρέσεις. Οι συμφωνίες για τον καθορισμό των τιμών ή μάλλον οι συμφωνίες για τις συμβάσεις οι οποίες θα υπογράφονται θα πρέπει να μην είναι υποχρεωτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης τιμών. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης και ένας ευρωπαϊκός κώδικας χρηστών πρακτικών όπως επίσης και ένα εθελοντικό πρόγραμμα Some πιστοποίησης των προϊόντων. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ε, επεκταθεί η χρήση τους γιατί βοηθούν τη σωστή στρατηγική της αγοράς και της οικονομίας κλίμακας. θα πρέπει να βελτιώσουμε τον συντονισμό ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Βέβαια η διαχείριση ε, των κρίσεων και η διαχείριση των κινδύνων μέχρι τώρα δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στις αντιδράσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα. Άδες άλλα μέτρα είναι τα μέτρα της αντιπροσώπευσης των γεωργών της επαγγελματικής τους εκπροσώπησης δηλαδή, η αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα και θα πρέπει να υπάρξει και ένας κεντρικός ρόλος στη σχεδίαση συμβολέων, συμβάσεων οι οποίες να είναι θα έλεγα σχετικά τυποποιημένες σχετικά με τον ανταγωνισμό θα πρέπει να ληφθούν και εκεί μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στην αγορά και με τα προηγούμενα μέσα και με νέα μέσα. Τώρα για τα σχολικά προγράμματα θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμός με τον τομέα της παραγωγής οπωροκυπευτικών και λαχανικών γενικότερα. Η βοήθεια σε κοινωνικά εύθραυτες ομάδες είναι ένας στόχος που έχει άμεση σχέση με την ανακούφιση από την φτώχεια. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους μηχανισμούς αύξησης της πρόσβασης σε προϊόντα τα οποία αντιμετωπίζουν κρίσεις και σοβαρά προβλήματα. Περνάμε τώρα σε, έναν άλλο, σε μια άλλη ομάδα αμέσων την διαχείριση κινδύνου. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες βασικές αρχές. Από τη μία υπάρχει ανάγκη για διαφοροποίηση της αντίληψης του κινδύνου στη γεωργία, ευέλικτα συναχρηματοδοτικά προγράμματα, κανένα μέσο δεν θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν, να υπάρχει κατανομή των κινδύνων και συνυπευθυνότητα, βελτίωση της εκπαίδευσης των γεωργών και της ενημέρωσής τους, και ε, κοινέ βασικές ε, νομικές ρυθμίσεις γύρω από την γεωργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν αυτό που ονόμασα προηγουμένως ένα μέσο εγγύησης των εισοδημάτων των γεωργών. Θα πρέπει να είναι από την πλευρά του δημοσίου, να προωθεί τη ε, υπευθυνοποίηση θα έλεγα όλων, να συνδυάζεται η χρηματοδότηση από όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτό σημαίνει ότι το μέσο αυτό θα πρέπει να έχει, ε, θα έλεγα να είναι συμβατό με το λεγόμενο πράσινο κουτί. Τα μέσα τα οποία προτείνουμε θα πρέπει να βασίζονται είτε σε κρατικές βοήθειες είτε στο άρθρο 68. Δίνω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου που θα συνεχίσει στην Ισπανική. Στα μέτρα αντίδρασης ε, περιλαμβάνονται τα παραδοσιακά μέσα, τα οποία, τα οποία ήδη γνωστά στην ε, γεωργική πολιτική, την ε, αποθήκευση κλπ. Στη μελέτη αναφέρουμε ότι το σύστημα της αποθήκευσης θα πρέπει να διατηρηθεί και ως έχει, να μην τροποποιηθεί δηλαδή, και σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία στα σύνορα υπάρχει κάποιο δυναμικό σύμφωνα με τις ε, δυνατότητες πρόβαση στην αγορά. Αυτό θα πρέπει, ο θα πρέπει να διατηρηθεί ιδιαίτερα σε περιπτώσει όπου οι τιμές είναι υψηλέ ε, στι πρώτε πρώτες ε, κάτι το οποίο ενδεχόμενα να απειλεί διαφορετικά την, τον εφοδιασμό τη κοινή αγορά. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχει δυνατότητα να μειώσουμε ή να καταργήσουμε του δάσμου Και κάτι ακόμα, ε, υπάρχουν δεσμεύσει ε, σε ό,τι αφορά τους εμπορικούς γύρους, ε, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγεί σε μείωση των δασμών και δημιουργεί κάποιες ε, αναταραχές στις αγορές σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ρήτρες προστασίας για ευαίσθητα προϊόντα τώρα. Ότι τη παραγωγή των προϊόντων αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί όπως, ε, όπως έχει και να αφορά τα προϊόντα υψηλής ε, πολιτικής αξίας όπως οι ονομασίες προέλευσης και όλες οι πολιτικές ε, για την υψηλή ποιότητα και για τα προϊόντα τα οποία έχουν συγκεκριμένα ε, συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες χαρακτηριστικά όπως τα οικολογικά προϊόντα κλπ. Επίσης, σε φορά την προαγωγή στον τομέα των απορροκυπευτικών και για τον τομέα του ίνου. Έχουμε εδώ κάποιες νέες δυνατότητες δράσης με την έννοια ότι υπάρχουν νέες επιπτώσεις όχι μόνο λόγω της, του ανοίγματο νέων αγορών αλλά διότι ενισχύουν και την αλυσίδα προμήθειας αυτών των προϊόντων. Ε, αναφέρομαι εδώ σε προϊόντα που αφορούν ε, τρίτες χώρες ε, και τέλος ε, στη μελέτη περιλαμβάνονται και οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων όπως σε περιπτώσεις όπου όλα τα υπόλοιπα μέσα απέτυχαν και δεν μπόρεσαν να ε, βελτιώσουν μια κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τις ε, ε, αποζημιώσεις επιπτώσεις καταστροφών ή και μέτρα τα έκτακτα όπως τα φορολογικά ή την πρόσβαση στον, στην πίστη με βάση τα εθνικά προγράμματα, τα εθνικά εθνιστικά προγράμματα. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα σε σοβαρών διαταραχών να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα και για να επιτραπεί κάτι τέτοιο πάντα προκειμένου για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων απρόβλεπτων θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός αποθέματος στον προϋπολογισμό θα είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων όταν έγινε η κατάρτιση των προπολογισμού. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα κλαδικό σύστημα. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα του, του βοήου κρέατος και την διαχείρισή του με τρόπο ολοκληρωμένο, ομοιογενή. Εντός των μέτρων διαχείρισης ε, των κρίσεων ε, θα υπάρχουν ε, τα αμοιβαία μία, τα προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την σωστή ενημέρωση προκειμένου να επιτρέψουν την ενσωμάτωση αυτών των μέτρων διαχείρισης ε, των ε, κρίσεων στον τομέα των, ε, του κρέατος και των κτηνοτροφικών. Δημιουργία συμβάσεων τύπου κάτι το οποίο θα επιτρέψει να μειωθούν οι αβεβαιότητες και η χρήση ε, βέλτιστων πρακτικών. Εάν δεν παρκέψουν αυτά τα μέτρα για την διόρθωση της κρίσης και την αντιμετωπισή της, θα μπορούσαμε να προσφύγουμε στο θέμα της δημόσιας ε, αποθήκευσης, ε, α, αποθεματοποίησης καλύτερα, όπως για τα δημητριακά, τα σιτηρά και την ε, ρήτρα προφύλαξης. Και φυσικά ε, πρέπει να γίνουν προσαρμογές ε, κατάλληλες για κάθε τομέα. Καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα εδώ, όπου τονίζουμε την αγιότητα να γίνουν προοδευτικές αλλαγές από ένα μοντέλο δημόσιας στήριξης σε ένα μοντέλο έμεσης δημόσιας στήριξης και μέτρα τα οποία θα επικεντρώνονται στην διαχείριση των κρίσεων. Η Γεωργία θα πρέπει να διαθέτει λοιπόν κοινού κανόνες που θα στηρίζουν ένα, μια ε, ισχυρή ε, αλυσίδα τροφίμων. Κάθε κλάδος έχει ανάγκη από δικά του πρωτόκολλα και τα μέτρα αυτά ως εκ τούτου χρειάζεται να αποδεσμεύονται μέσω των ρυθμίσεων των τιμών. Η διαχείριση των κρίσεων θα πρέπει μάλλον την ε, μέτρα θα λαμβάνουν όπως καταλαβαίνετε μετά από την εκδήλωση της κρίσης. Τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει στην ε, καλύτερη διαχείριση των ε, διεθνών αγορών μέσω της διαφάνειας και της ενημέρωσης και τους καλύτερους συντονισμούς με άλλες ε, κοινέ πολιτικές που, όπως η εμπορική πολιτική, η οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική κλπ. Αυτά ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε τους ε, εισηγητές μας. Να ξεκινήσουμε σε μέρος τη συζήτηση. Ακούσαμε ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις. Ε, θα ξεκινήσουμε με τον Έλμπερτ Ντόφμαν. Έχεις το λόγο, Έλμπερτ. Και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όντως είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα των οργανώσεων οργανάς αγοράς είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει μέσα από τη μεταρρύθμιση της ε, γεωργικής ε, πολιτικής που συχνά λησμονείται και όμως έχει κεντρικό χαρακτήρα και σημασία. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό το τι έχουμε αυτή τη μελέτη και εγκαίρως. Και μη τι άλλο θα πρέπει οι μηχανισμοί αγοράς που υφίστανται ακόμη, κάποιες κοινέ οργανώσεις αγοράς επίση που παραμένουν, δεν θα πρέπει να λησμονηθούν. Γιατί πιστεύω ότι τις χρειαζόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως θετικό το παράδειγμα των απορολαχανικών όντως, η τροποποίηση της κοινή οργάνωση αγοράς των απορολαχανικών το 1996 οδήγησε όντως σε μια θετική εξέλιξη για την αγορά, ε, καλύτερη οργάνωση, άνοιγμα της αγοράς και γι' αυτό πιστεύω ότι το πρότυπο αυτό, τα λειτουργικά δηλαδή προγράμματα, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο σύστημα και σε άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει να, μας, το δούμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης τώρα. Αυτό ίσως σε σχέση με τις προτάσεις που γίνονται για το συνεταιρισμό. Δεύτερον, είναι όντως σημαντικό και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει να παρουσιάσει προϊόντα ε, μεταποιημένα ύψης της ποιότητας που έχουν καλές ευκαιρίες για παρουσία και αξιοποίηση στις ε, διεθνείς αγορές. Νομίζω λοιπόν και μάλιστα υπάρχει και οριζόντιος κανονισμός ε, για την εκστρατεία, τη διαφημιστική ή την επικοινωνιακή καλύτερα για τα προϊόντα αυτά. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι αυτός ο κανονισμός δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση για την σχετική εκστρατεία και δεύτερον το σύστημα και το πρότυπο το οποίο ακολουθείτε οδηγεί τελικά στο να μην ενδιαφέρονται οι επιχειρήσει να συμμετάσχουν σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωση. Γιατί δεν εξασφαλίζονται καλύτερε προσβάσει στι αγορέ. Εάν, ε, παραδείγματι, μια, αγορά έχει, μια επιχείρηση έχει να προβάλλει ε, γάλα, κρέας, λαχανικά, ό,τι είναι από την ευρωπαϊκή παραγωγή, δεν έχει τίποτε συγκεκριμένο να αποκομίσει και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία. Έτσι λοιπόν με τον οριζόντιο τύπο του κανονισμού, νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και επικοινωνιακά την ευρωπαϊκή παραγωγή. Έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις μας να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία αυτή και να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ε, διέξοδο στις αγορές για τα προϊόντα τους. Εάν χρειάζεται και με τη συγχρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μελέτη νομίζω αξίζει να αναλυθεί διεξοδικότατα, ειδικά τώρα που ε, πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της διαμόρφωσης της γεωργικής πολιτικής μετά το 2013, θα πρέπει να δούμε τι προκύπτει ως αποτέλεσμα, ως σύσταση από αυτή τη μελέτη. Διότι εγώ βλέπω ότι ως προς τα προβλήματα τα σχετικά με την παρέμβαση δεν βλέπω να γίνεται αρκετό λόγο εδώ. Και όμω έχουμε πολλέ δυσκολίε με το 2000. Θα έχουμε μάλλον πολλέ δυσκολίε με το 2013 για τα θέματα τη παρέμβαση. Και καλό θα, πρέπει, θα είναι να τα εξετάσουμε. Τα δίκτυα ασφαλείας. Αυτά θα πρέπει να ε, καλύψουν και τον καταναλωτή όπως και τον παραγωγό. Δηλαδή να υπάρχει και προστασία του εισοδήματο του παραγωγού αλλά και αδιασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλούμε για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, πολιτικής, της γεωργικής πολιτικής που είναι η παρέμβαση και εδώ θα αναφερθώ καλύτερα, ε, πιο συγκεκριμένα στα σιτηρά, στην αγορά των σιτηρών που θεωρώ πολύ σημαντική γι' αυτό και την επαναλαμβάνω διαρκώς. Ε, τι πρόβλημα έχουμε προς τη χρηματοδότηση εδώ. Έχουμε αναπτύξει διάφορες δομές, έχουμε δομές και στη τραπεζικό τομέα και στα χρηματιστήρια. Χρειάζεται λοιπόν και στον τομέα της γεωργίας η δομή της επιτήρησης. Επιτήρηση για να έχουμε αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες, για ε, να μπορούμε και τις σωστές αποφάσεις να λαμβάνουμε δεδομένες ε, της ε, αλλά και να αντιμετωπίσουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα της γεωργικής πολιτικής. Επίσης, τα διάφορα διδάγματα που μας έχει προσφέρει η εμπειρία μας από το παρελθόν και από την παρέμβαση ιδιαίτερως, θα πρέπει να τα συλλέξουμε και να τα συναγάγουμε και βέβαια με αξιολόγηση κινδύνου, αλλά και με εκτίμηση κόστους συγκεκριμένα. Μια και έγινε λόγος γι' αυτό δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι δομές οι οποίες θα συμμετάσχουν, φερειπίν μέσω του παραγωγού ή ε, εάν θα έχουμε διαφορετικές δομές. Επίσης, η επιστηστική βοήθεια για τους φτωχούς ε, πολίτες ή για τα παιδιά που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια θεωρούνται μέτρα γιατί εξυπηρετούν κάποιους συγκεκριμένου στόχους της αγοράς ή μπορεί να επιδιώκουν κάποιον άλλον στόχο, φερρυπίν, βελτίωση της δημόσιας υγείας, και ούτω καθεξής. Γιατί ξέρουμε ότι τέτοιου είδους μέτρα ε, συχνά παρουσιάζουν το φαινόμενο της επικάλυψης της τομεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή η γεωργική πολιτική, είναι και κοινωνική πολιτική. Αφόσον προσφέρεται βοήθεια στη διατροφή ή επιστηστική βοήθεια. Άρα θα πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα αυτή η επιστηστική βοήθεια για φτωχού και για παιδιά που υπάγεται. Είναι και τεράστια σημασία αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Μια ερώτηση μόνο. Γιατί ακούγεται ο όρος συνέχεια ασφάλιση ως στοιχείο στήριξης της αγοράς σε αυτές τις παρεμβάσεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να εμποδίσουμε αυτά τα χρήματα της στήριξης ε, για τη γεωργία ε, να μην καταλήγουν, να καταλήγουν στην ε, ε, ασφάλιση τελικά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι τα αξιοποιεί ο παραγωγός για προσωπικό κέρδος και όχι για το σκοπό για τον οποίο έχει προβλεφθεί. Έτσι λοιπόν πρέπει να του πούμε ότι ναι, θα έχεις και τη στήριξή σου και θέλουμε να δούμε τι ασφάλιση θα συνάψει και ότι τα χρήματα αυτής της στήριξη θα πάνε αποδεδειγμένα, φερειπίν στην αγορά καινούριων μηχανήματος ε, και ούτω καθεξής. Ε, είναι ένα σύστημα το οποίο φοβούμε ότι θα ε, μεταφερθεί ως έχει στην ασφάλιση. Και πρέπει οτιδήποτε προβλεφθεί στην υπόθεση αυτή να είναι απόλυτα ασφαλές, να μην υπάρχουν παραθυράκια για κατάχρηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χόισλινγκ για, ε, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσαν οι ομιλητές. Ακούσαμε και τη σπάνιο γεγονός ότι η λέξη καταναλωτής είναι από τις λίγες περιπτώσεις που σε μελέτες ακούγεται ο όρος καταναλωτής και αξιοποίηση από την αγορά. Εν πάση περιπτώσει παραμένουν πολλά ερωτηματικά για το πώς προσδιορίζεται παραδείγματι το όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου Η αποθεματοποίηση επίσης ε, πάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού ε, τομέα, γιατί αυτό το ζήτημα των αποθεμάτων έχει πολύ μεγάλη σημασία για την καθοδήγηση των αγορών και είναι χρήσιμο εργαλείο. Ένα πράγμα το οποίο δεν είδα να αναφέρεται παρκώς στις παρουσιάσεις ήταν η διαφάνεια και η επιτήρηση των αγορών. Αυτό που λέμε monitoring για το τι σημαίνει ε, για το τι συμβαίνει στι αγορές, που αποτελεί βέβαια και προϋπόθεση της ε, διαφάνεια. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, προσοχή στη διαφάνεια και την επιτήρηση των αγορών και δεν θέλω περισσότερη έμφαση. Εμείς όπως και οι φιλελεύθεροι συμφωνούμε στο θέμα της ε, ασφάλισης. Έχω πολλές επιφυλάξεις ε, γιατί εδώ πάλι έχουμε ε, επικαλύψει μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καλό θα είναι να μην υποστηρίζει με κονδυλιά του ο δημόσιος τομέας την ιδιωτική ασφάλιση. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό αυτό και θα πρέπει να δούμε πού καταλήγουν τα χρήματα. Αυτά φυσικά θα χρειαστεί να το συστήσουμε διεξοδικά. Και άλλη μια ερώτηση, όταν γίνεται λόγος για δίκτυα ασφαλείας. Το σημαντικό ερώτημα είναι ποιο θέτει σε λειτουργία αυτό το μηχανισμό ασφαλεία και πότε, υπό ποιου όρου. Το είδαμε και με την κρίση στα γαλακτοκομικά. Ότι ετέθη σε λειτουργία ένα μηχανισμό ο οποίο μπόρεσε να ενεργοποιηθεί 1,5 χρόνο μόλις αφού είχαν περάσει 1,5 χρόνο η γαλακτοπαραγωγή πουλώντας το γάλα τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Άρα χρειαζόμαστε πιο γρήγορους μηχανισμούς. Ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Okay. Και ευχαριστώ τους συντάκτες των μελετών. Βλέπω με χαρά ότι υπάρχει ευρύτερη συνένεση στα θέματα που επισημαίνουν οι συνάδελφοι, κάτι που θα χρειαστούμε και στο μέλλον για την αναθεώρηση ορική πολιτική, γιατί βεβαίω πρώτο μέλημα θα πρέπει να είναι η ε, προμήθεια σε τρόφιμα για τον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά ταυτόχρονα και η στήριξη τη γεωργία και του παραγωγού μα. Γιατί του χρειαζόμαστε του παραγωγού. Πολλά είναι τα ερωτηματικά. Ακούστηκαν αρκετά νωρίτερα. Εγώ έχω τέσσερα να διατυπώσω. Πρώτον, για να καταλάβω καλύτερα τις προτάσεις, ε, μιλήσατε για μέσα ρύθμισης της αγοράς που θα λειτουργούν είτε, θα, θα προβλέπονται είτε για κάποια ομαλώς λειτουργούσα αγορά, είτε σε άλλη περίπτωση για αγορά που αντιμετωπίζει κρίση. Τι σημαίνει όμως ομαλώς λειτουργούσα αγορά. Πώς θα οριστεί τα μέσα αυτά ρύθμιση αγοράς θα είναι στα χέρια περισσότερο των παραγωγών του κλάδου. Εγώ θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτική θα πρέπει πάντοτε να παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση κρίσης, όπου υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες μιας κρίσης. Καλά το κατάλαβα και αυτό ακριβώς έχετε προτείνει κάτι διαφορετικό. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα πρέπει σε ομαλές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς να παρεμβαίνει παρόλα αυτό το κράτος. Δεύτερη ερώτηση. Έχετε κάποια ιδέα συγκεκριμένη να προτείνετε ως προς την αντιμετώπιση το, της κερδοσκοπίας στην αγορά, ως εκ τούτου της κερδοσκοπίας στις τιμές. Γιατί φαντάζομαι βέβαια ότι θα ενθουσιαστεί ο οποίο παραγωγός να ε, εκτοξεύονται οι αγορές στα ύψη. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει πάντοτε παράλληλα για όλα τα προϊόντα. Ε, αν ανέβει η τιμή στα στηρά, μπορεί να πέφτει φερρυπή τα γαλακτοκομικά και άρα πότε ο ένα αισθάνεται ικανοποιημένο και πότε ο άλλο. Αυτό πώ θα το ε, συζητήσουμε, πώ θα το αντιμετωπίσουμε μέσα από τις ε, οργανώσεις αγοράς. Τρίτον, πώς βλέπετε και πώς ορίζετε εσείς τη σχέση μεταξύ της ιδιωτικής ευθύνη και πρόληψη ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων από πλευρά του παραγωγού και της παρέμβαση από την αγορά. Και αυτό το λέω διότι στην περιοχή μου όταν είχαμε τις εγγυήσεις τιμών για τον παραγωγό. Δεν μπορέσαμε να τον σώσουμε τους παραγωγούς όταν πράγματα, τα, πράγματα πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας την εποχή εκείνη. Δεν μπόρεσε να σώσει τους παραγωγούς, δεν, μπορούσε, δεν μπορούσε καν να σωθεί το ίδιο το κράτος γιατί χρεοκόπησε. Ε, άλλη ερώτηση σχετικά με την παρέμβαση επιστροφές εξαγωγών για το μέλλον είναι ένα μέτρο το οποίο θεωρείτε ότι μπορεί να διδραματίσει κάποιο ρόλο ή όχι. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι ήταν σημαντικές οι παρεμβάσεις σα, Όλοι ανησυχούμε για το πώς θα λειτουργήσει η καινούργια αυτή ΚΑΠ από το 2013 και κατά πόσο θα είναι καινοτόμο στους τρόπους διαχείρισης των κρίσεων σαν και αυτό που ζήσαμε στο γαλακτοκομικό τομέα. Ξαναδίνω το λόγο στους δύο εισηγητές λοιπόν για να δώσουν απαντήσεις και περνάμε μετά στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Ξεκινώντας από τις τελευταίες ερωτήσεις τι γνώμη έχουμε για τις επιδοτήσεις των εξαγωγών. Ε, η Μερέτη αποφάνθηκε υπέρ της ε, κατάργησης. Θεωρούμε ότι δεν είναι αποτελεσματικός μηχανισμός για να διαχειριστούμε τις ε, αγροτικές, τις γεωργικές αγορές. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευθύνη του Γεωργού κλπ. Νομίζω ότι τα ισχύοντα μέτρα επαρκούν για την τήρηση των ελάχιστων τιμών. Τώρα η κερδοσκοπία νομίζω ότι είναι η κερδοσκοπία των ε, χρηματαγορών. Ε, προσπάθησα να το συμπεριλάβω αυτό στις, ε, στα συμπεράσματα, δηλαδή να υπάρχει καλύτερη πειθαρχία στα, αγορέ αγορές παραγόγων. Είναι απαραίτητη η παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων. Θα ήθελα να απαντήσω την ερώτηση που τέθηκε για το γαλακτοκομικό τομέα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις καταστάσεις κρίσης και ότι η πολιτική μας έχει μετακινηθεί και έχει ε, μεταφερθεί σε μια έμεση στήριξη προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικότερα οι αγορές. Η φυσιολογική κατάσταση λοιπόν ε, θα πρέπει να οδηγήσει σε μια καλύτερη πειθαρχία μέσω ενίσχυσης των μηχανισμών που ε, καθορίζουν και διέπουν ε, την αλυσίδα των, τιμών. Αυτό συνέβη και με το γάλα. Στην αρχή χρειάστηκε να αντιδράσουμε άμεσα, οι αγορές δεν ήταν διάφανες και υπήρξε μεγαλύτερη, ιδιαίτερη ανισορροπία σε επίπεδο τιμών. Θεωρούμε λοιπόν ότι η γεωργική πολιτική θα πρέπει να ε, επιδρά περισσότερο για τη δημιουργία ενό πλαισίου το οποίο αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι σχέσει των γεωργών με του υπολείπου εμπλεκόμενου των αλυσίδα και στον κλάδο. Επίση ε, θα ήθελα να πω ότι ε, υπόθηκαν κάποια σχόλια με τα οποία, για τα οποία είμαστε υπέρ τουλάχιστον η δυνατότητα επέκτασης των ε, προγραμμάτων των απορριφτικών και σε άλλους τομείς, ιδιαίτερα για τα διαφορετικά προϊόντα όπως τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και κρίνουμε ότι η αγροτική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στους καταναλωτέ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευστική βοήθεια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή μας την παρουσίαση. Να δώσω λόγο στον Αλμπέρτο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω την ερώτηση. Το σχετικό με το ρόλο του ιδιωτικού και του ε, δημόσιου τομέα στα μέσα διαχείρισης κινδύνων και ασφάλιση. Προτείνουμε εμείς μια βασική κάλυψη. Αυτή η βασική κάλυψη δημιουργεί ένα δίκτυο προστασίας στο σύνολο των πιστώσεων, όχι σε ένα συγκεκριμένο τομέα για μια συγκεκριμένη παραγωγή. Υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή ασφαλιστικές συμβάσεις που προσφέρονται προς τους γεωργούς από τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προτείνουμε λοιπόν αυτό το δίκτυο προστασίας να μην προτείνεται, να μην προσφέρεται δωρεάν, αλλά να υπάρχει μια βασική κάλυψη έτσι ώστε να ε, υπευθυνοποιούνται οι γεωργοί και ταυτόχρονα να προσφέρει αντίστοιχα ποσά και πιστώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σωστή λειτουργία του δικτύου προστασίας, ένα δίκτυο προστασίας το οποίο θα είναι συνδυασμός ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δεν προτείνουμε εμείς να δοθούν επιπλέον επιδοτήσεις σαν ασφάλιση προς τους γεωργούς. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε τα βασικά των βασικών στα πλαίσια ενός συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Μπαντάζη και τον κύριο Γκαρίντο για την παρουσίασή τους και για τη συζήτηση που ακολούθησε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν ζητήσει το λόγο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης τροποποίηση του κανονισμού 7309 του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τα καθεστώτα στήριξης, άμεσης στήριξης στους γεωργούς. Έχουμε δύο πακέτα ουσιαστικά για την ευθυγράμμισή μας με τη Λισαβόνα. Όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, Ήμασταν ιδιαίτερα δραστήριοι ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προσαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας το ταχύτερο δυνατόν στις νέες προβλέψεις ε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνα σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και στην Επιτροπολογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον Τάτσι Τσόλος που θα έχουμε αύριο εδώ για την ταχύτητα με την οποία παρουσίασε τις προτάσεις αυτές προσαρμογής. Αυτές που θα εξετάσουμε σήμερα είναι οι δύο πρώτες, αλλά θα υπάρξουν αρκετές δεκάδες πακέτα νομοθετικών αλλαγών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα λοιπόν το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια αυτού του πακέτου άμεσης βοήθειας προς τους διαργούς που απαιτούν αλλαγή του κανονισμού 73-2009. Σαν εισηγητής εγώ θέλησα να εισάγω ορισμένε τροποποιήσεις σχετικά με την πρόταση την οποία έκανε για την προσαρμογή και ευθυγράμμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνω υπόψη το λεγόμενο common understanding ανάμεσα στα όργανα και τον κανονισμό σχετικά με τις εκτελεστικές πράξεις. Θεωρώ ότι όταν πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις στην βασική πράξη, ή όταν αντιμετωπίζονται τα θέματα των δικαίων των γεωργών θα πρέπει αυτό να γίνεται μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Πράξεων δηλαδή τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να μπλοκάρει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω απλών εκτελεστικών πράξεων ή μέσω πράξεων για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης. Θεωρώ επίσης απαραίτητη να υπάρξει μια τροποποίηση του άρθρου 11 του κανονισμού στα πλαίσια του οποίου το Συμβούλιο, το Συμβούλιο επαναλαμβάνω, έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία. Στο συγκεκριμένο σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει κάποια πρόταση τροποποίησης και αφήνει ως έχει μια ρύθμιση η οποία είναι θα έλεγα ασύμβατη με τη σημερινή νομοθετική πραγματικότητα μετά τη Λισαβόνα στα πλαίσια της οποίας ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει ομότιμα στην διαδικασία την ομοθετική που αφορά και την κοινή αγροτική πολιτική και το προϋπολογισμό συνολικά της Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνω μέσω της τροπολογίας 7 να υπάρξει μια τροποποίηση έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δημοσιονομική πειθαρχία λαμβάνοντας υπόψη α, τους σύντομους χρόνους μέσα στους οποίους θα εξελιχθεί η μέθοδος αυτή. Αυτά ήταν τα σημαντικά τώρα για τις προτάσεις απλοποίησης που εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να εισάγουμε κάποια επιπλέον στοιχεία ευελιξίας και απλοποίησης για την ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού από πλευράς όλων των κρατών μελών. Όπως πάντα, εγώ θα ακούσω προσεκτικά τις παρατηρήσεις σας, θα λάβω υπόψη τις τροπολογίες σας και θα πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία με το Συμβούλιο και να στείλουμε λοιπόν ένα γρήγορο μήνυμα για την πραγματική μας βούληση να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό της ευθυγράμμισης με τη νέα συνθήκη. Ε, δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι εμείς είμαστε η πρώτη κοινοβουλευτική επιτροπή χάρη στον Επίτροπο Τσιόλος η οποία παράγει νομοθετικές πράκτης ευθυγράμμισης με τη νέα συνθήκη. Κλείνοντα θα ήθελα να ερμηνεύσω το πνεύμα της Επιτροπής μας λέγοντας ότι όλοι έχουμε την επιθυμία να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις νέες ρήτρε τη συνθήκη, οι οποίες προβλέπουν μια πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίασή μου. Τώρα θα δώσω το λόγο πρώτα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, για μια στιγμή. Πρώτα οι συνάδελφοι που θα ζητήσουν το λόγο. Πρώτα οι συνάδελφοι. Μάιερ, πρέγω. Εκ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Άλντε. Υποστηρίζουμε τις ε, προτεραιότητές σας τις δικές σας και βέβαια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πάολο. Πολύ καλή έκθεσή σου, πιστεύω. και διέκρινες ιδιαίτερα πολύ καλά μεταξύ των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών διατάξεων πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να το δούμε αυτό το θέμα. Είναι αυτό το οποίο μπορέσαμε χάρη σε χρόνους αγώνων να επιτύχουμε. Έχουμε δηλαδή ξεφύγει από το παλιό σύστημα της επιτροπολογίας και μπορούμε εμείς να παρεμβαίνουμε και να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματά μας ε, στη νομοθετική διαδικασία και έτσι δεν ε, εκχωρούμε εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλώς μπορούμε να επιταχύνουμε την νομοπαραγωγική διαδικασία διαφυλάσσοντας όμως τον δικό μας, ε, τη δική μας παρέμβαση μέσα από ένα μηχανισμό ελέγχου ε, σε περίπτωση που πρόκειται για νομοθετική διαδικασία και όχι για απλή τεχνική προσαρμογή. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο για τις ε, τροπολογίες που θα καταθέσουμε και που θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες, τα επιμέρους σημεία. Ως προς το περιεχόμενο δεν έχουμε ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερες παρατηρήσεις, μόνο στην απλούστευση θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερα στις κατεξουσιοδότηση ε, πράξης όπου θα θέλαμε τη διατύπωση κατά τρόπον ώστε να διαφυλάσσονται τα δικαιώματά μας και να γίνεται βέβαια και πιο απλός ο τρόπος παραγωγής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπερθυμίζω ότι στι 22 Μαρτίου στι 12 το μεσημέρι είναι η καταληκτή υποθεσμένη τροπολογιών. Αν θέλει κάποιο συνάδελφο ε, να υποβάλει τροπολογία. Ο Λεμίτσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την έκθεσή σου. Είναι πραγματικά πολύ καλή. Και σε ό,τι αφορά τώρα την προσαρμογή στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που ενδεχόμενα να πρέπει να συζητηθούν ενδελεχέστερα αλλά έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά με την απλοποίηση της ε, ΚΑΠ και θα υποβάλω ανθρωπολογίες περί αυτού. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε επανειλημμένα ότι αυτή η απλοποίηση θα σημαίνει καλή τη λειτουργία στην πράξη των ε, θεσμών. Και δεν βλέπω όμως να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση εδώ, π.χ. στο ζήτημα της πολλαπλής συμμόρφωσης ε, ή και στο ζήτημα των ελέγχων. Εάν ε, κατάλαβα καλά, εμείς δεν είμαστε υπέρ του αύξηση του διοικητικού άχθους των ελέγχων, εάν η αμέλεια είναι ίσονος ε, σημασίας. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε λίγο παραπάνω το ζήτημα της απλοποίησης και των ελέγχων. Ευχαριστώ. Ζωζέ Μποβέ. Έχεις το Ναι. Κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με το ότι το ζήτημα αυτό προχώρησε εντάχει. Ίσως θα έπρεπε να γίνει μια συλλογική δουλειά προηγούμενα θα ήταν σημαντικό προτού να υποβληθούν οι προτάσεις ε, ίσως λοιπόν σε επίπεδο μεθοδολογίας ε, θα έπρεπε να έχουμε μια συνάντηση με το σύνολο των πολιτικών ομάδων για να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε αποτελεσματικότερα. <clears throat> Διότι, όπως υπενθυμίσατε, ήμασταν η πρώτη επιτροπή που δούλεψε προκειμένου να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της δίκης αγώνας. Και αυτό με οδηγεί στο διαρωτηθώ επί δύο τροπολογιών, τις οποίες δεν καταλαβαίνω. Τροπολογία επαρχήμων 3 είναι η πρώτη, όπου αφαιρούμε ένα μικρό κομμάτι και καμία ενίσχυση δεν γίνεται προς τους παραγωγούς. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί μιλάμε για τη ε, δημοδότηση των ε, φυλαζουσών αγελάδων και τροπολογία 12 Ήδη ίδια η διατύπωση του τροπολογία 12 μου είναι απολύτω ακατανόητη. Θα ήθελα λοιπόν κάποιε εξηγήσει, διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώ παίζεται. Ωραία. Λουίς Κάπουλας Σαντόζα. Παρακαλώ, Λουίς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να πω ότι από πλευρά τη σοσιαλιστικής ομάδας. Εμεί υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Επιτροπής. Εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, την προσπάθεια για διαφύλαξη των ε, προνομιών και εξουσιών του Κοινοβουλίου με την ορθή εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Σε ευχαριστώ, Λουί. Πρωτού να δώσω το λίγο στον ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζω την καρλική ημερομηνία 22 Μαρτίου. Υπενθυμίζω στους συναδέλφου ότι πρόκειται για μια προσαρμογή της νομοθεσίας στη συνθήκη της Λισαβόνα. Ω εκ τούτου, εμεί χρειάζεται να δουλέψουμε επί των ζητημάτων που άπτονται των κατευθυντών πράξεων και τη εκτελεστική πράξη δεν πρόκειται να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις ε, θα τις κάνουμε με συνεννόηση με τις άλλες ε, ομάδες. Εκτός από κάποια απλοποίηση, κάποια αναδιατύπωση, αν θέλετε, του κειμένου. Εμείς να δώσω ευθύ αμέσως το λόγο στην κυρία Πατσέκο, στον κύριο Πατσέκο, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας, για τη δική μας πρόταση σχετικά με τη ρύθμιση των άμεσων βοηθειών, σύμφωνα πλέον με τη νέα συνθήκη. Χαίρομαι γιατί και εσείς κύριε Πρόεδρε και οι εισηγητές ε, υποστηρίζουν την πρόταση την οποία έχουμε κάνει στο σύνολό της. Διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα υψηλότερο ποσοστό σύγκλησης ανάμεσα στο δικό σας σχέδιο εκθέσεως και σε αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς. Να μου επιτρέψετε εδώ να σας μεταφέρω και τις πρώτες μας αντιδράσεις στις τροπολογίες σας. Τροπολογίες ελπίζω να φανούν χρήσιμες. Θα κάνω εδώ μια κάποια διάκριση ορισμένων θεσμικών θα έλεγα, ανάμεσα σε ορισμένες θεσμικές τροπολογίες και στις οποίες έχουμε αφήσει κενό και για τις οποίες δεν υπάρχει καμία δυσκολία θα κάνουμε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ε, για τον, ε, από τον κανονισμό για τη νέα επιτροπολογία και για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Υπάρχουν επίσης οι τροπολογίες συντακτικής φύσεως, οι οποίες δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν όμως τρία είδη τροπολογιών, πάνω στις οποίες θα ήθελα να επεκταθώ λίγο. Οι πρώτες τροπολογίες είναι αυτές οι οποίες κατά τη γνώμη μας προϋποθέτουν ορισμένες αλλαγές επί της ουσίας. Ε, οι 12, 14 και 16 σαν παράδειγμα. Όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παραμείνει στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης ανάμεσα στο τι υπάρχει με τη νέα συνθήκη δεν προχωρήσαμε και δεν προτείναμε κάποιες αλλαγές επί της ουσίας. Τώρα θα μπω αν θέλετε στην ουσία της συζήτησης για τις υπόλοιπες τροπολογίες οι οποίες ε, θα έλεγα ζητούν να υπάρξει τροποποίηση των εκτελεστικών πράξεων σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Να σας θυμίσω την μέθοδό μας, το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Για τις εκτελεστικές αυτές πράξεις θεωρήσαμε ότι είναι πράξεις που έχουν σαν μοναδικό στόχο να θέσουν σαν λειτουργία με ενιαίο τρόπο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει καθορίσει ο νομοθέτης. Οι εκτελεστικές πράξεις αντίθετα από τις πράξεις εξουσιοδότηση δεν έχουν σαν στόχο να τροποποιήσουν τις βασικές νομικές ρυθμίσεις. Είναι πράξεις για τις οποίες εμείς τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε τα δεδομένα τα οποία απλά μας έχουν δοθεί και απλά εκτελούμε ε, τις πράξεις αυτές σύμφωνα με τις αρμοδιότητές μας. Πέραν αυτού αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν παραρτήματα του βασικού κανονισμού. Εκεί πρόκειται για συγκεκριμένες τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν όλες τις αριθμητικές παρεμβάσεις που δεν αφήνουν καμία δυνατότητα αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να εμείνουμε στο πλαίσιο το οποίο μας καθορίζει η βασική ρύθμιση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση η οποία είναι ειδικού χαρακτήρα αφορά τα κατεπήγοντα μέτρα, το τροπολογία 9. Και εδώ έχουμε επιλέξει, αν θέλετε, τις, ε, τις εκτελεστικές πράξεις όπως προβλέπει ο κανονισμός. Θελήσαμε εμείς στα μέτρα του δυνατού να διατηρήσουμε το ε, υπάρχον καθεστώς. Αυτό τεκμηριώνεται νομίζω από την προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ταχύτατη, τη δυνατή αντίδραση σε κατεπίγουσες περιπτώσεις και σε περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια εκτελεστική πράξη λοιπόν η οποία τεκμηριώνεται από τον έκτακτο και ε, την χαρακτήρα της και την μεγάλη ανάγκη γρήγορης αντίδρασης. Μετά για την τροπολογία 7, Πρόεδρε, ζητάτε να αλλάξει η διαδικασία η σχετική με την διαδικασία που προβλέπεται σήμερα στον κανονισμό. Εδώ έχουμε προτείνει εμείς να κρατήσουμε τις αρμοδιότητες όπως προβλέποντο, γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για μια περίπτωση στην οποία το Συμβούλιο δεν λειτουργεί σαν νομοθέτης, αλλά αντιδρά χωρίς περιθώριο δράσης σε δημοσιονομικές συνθήκες οι οποίες προκαθορίζονται ουσιαστικά. Δεν υπάρχει λοιπόν ουσιαστικό περιθώριο δράσης από πλευράς του Συμβουλίου. Απλά το Συμβούλιο απαιτείται να λάβει υπόψη τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει από πριν. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας διαδικασίας ευθυγράμμισης, εδώ το συγκεκριμένο πλαίσιο ε, ε, προσφέρεται για περαιτέρω αλλαγές σε βάθος. Ε, τελειώνοντας Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι είμαι βέβαιος ότι οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και από τις δικές σας υπηρεσίες και από τις υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα συμβατό με τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει και αυτό σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ τον κύριο Πατσέκο τον ευχαριστώ για την παρουσίασή του. Είναι προφανές ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε τις λήψεις των αποφάσεων. Η ταχύτητα για μας, ταχύτητα αντίδρασης είναι κάτι το απαραίτητο, εφόσον όμως δεν είναι αντίθετη με τα δικαία τα οποία έχει το Κοινοβούλιο. Το κομβικό σημείο εδώ, πάνω στο οποίο ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, είναι εδώ εμείς λέμε ότι στις περιπτώσεις όπου ε, γίνονται κάποιες δυνατότητες στο Συμβούλιο παρέμβασης θα πρέπει να δίδονται και στο Κοινοβούλιο. Γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχουν διαφορές στις αρμοδιότητές τους. Συνεπώς εφόσον στο άρθρο 7 το Συμβούλιο δεν έχει περισσόριο δράσης, ανάλογα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται χωρίς περισσόριο δράσης βέβαια, αλλά δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Αυτό για μας είναι κάτι το απαράδεκτο και πρέπει να υπάρξει μια σαφέστατη και πιστή εφαρμογή στο πνεύμα και στο γράμμα της συνθήκης. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα δούμε σε επιμέρους επαφές πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θυμίζω τους συναδέλφους, τους συναδέλφους, ότι σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 73 του 2009, καθεστώς άμεσης στήριξης, η κατάθεση των τροπολογιών είναι η 21η Μαρτίου 12η μεσημβρινή. Ελπίζω να συμφωνήσετε για να προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού 1628 του 2005, δηλαδή στήριξη της ε, <clears throat> αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης και εδώ πρόκειται για προσαρμογή στην συνθήκη Λισαβόνας για την ε, αγροτική ανάπτυξη. Εδώ μιλάμε για έναν από του βασικότερου κανονισμού, Αυτό το 1698-2005. Η πρότασή τη η Κομισιόν ταξινόμησε τι περιπτώσει οι οποίε επιτρέπουν την υιοθέτηση ε, πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 τη συνθήκη. Δηλαδή, πράξεις γενικής φύσης, γενικού χαρακτήρα που τροποποιούν μη ουσιώδη τμήματα του κανονισμού αλλά και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τεχνικά στοιχεία και διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση, θα ήθελα να πω στους εκπροσώπους της Κομισιόν ότι σύμφωνο με την κατανομή που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τροπή και θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε σε αυτή την πρόταση να καταθέσω τροπολογία σχετικά με την ταξινόμηση ε, πράξεων και εκτελεστικών πράξεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτάσεις της Κομισιόν σε άλλες πτυχέ του κανονισμού, θεώρησα χρήσιμο να συμπεριλάβω κάποια στοιχεία από ε, πλούστευσης, ε, απλοποίησης και μεγαλύτερης ευελιξίας για να επιτρέψω την καλύτερη εφαρμογή της, ε, του κανονισμού. Οι υπόλοιπε τροπολογίε είναι οριζόντιου χαρακτήρα και τεχνικού χαρακτήρα και θα συμπεριληφθούν σε όλε τι προτάσει ευθυγράμμιση, διότι αντικατοπτρίζουν την κοινή στάση του Συμβουλίου και, της, και του Κοινοβουλίου στο θέμα των κατεξουδότηση πράξεων. Λοιπόν, ε, πάνω στο ζήτημα αυτό δεν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά απευθύνομαι και προς τους συναδέλφους και τους ερωτώ αν ε, έχουν ε, κάποιες προτάσεις, κάποια σχόλια να κάνουν. Παρακαλώ, συνάδελφοι, έχετε να προσθέσετε κάτι πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Πατσέκο. πριν να δώσω, όχι τον κύριο Πατσέκο, τον κύριο Σουζούβα. Λοιπόν, πριν να δώσω με το λόγο στον κύριο Σουσούβα. Δεν βλέπω οι συνάδελφοι να επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ο Διευθυντής κύριος Σουσούβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας και την διασαφήνιση αυτών των προτάσεων της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Διατηρούμε λοιπόν την ιδέα αυτή της ε, πράξης ε, ευθυγράμμισης και τη διάκριση μεταξύ κατεξουδότηξης πράξεων και εκτελεστικών. Όσον όμως αφορά τις οχτώ τροπολογίες σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι παριθμών 1, 2, 7 και 8 είναι όντως τροπολογίες οριζόντιου χαρακτήρα, θεσμικού χαρακτήρα. και με κείμενο σύμφωνο με το, με το Common Understanding, το κοινό μνημόνιο που αναφέρεται στην επιτροπολογία, η ΔΕ υπαριθμών 4 προβαίνει σε μια διευκρίνηση για την οποία δεν έχουν αντίρρηση οι υπηρεσίε επιτροπή. Μπορούμε να ακολουθήσουμε δηλαδή τη δική σα διατύπωση. Πλην όμω, διατυπώνω επιφυλάξει ω προ τι τροπολογίε 3, 5 και 6 όπου δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την δική σας επιχειρηματολογία. Συγκεκριμένα για την τροπολογία υπαριθμών 3. Τι έχουμε, να κάνουμε, τι έχουμε να δούμε εδώ. Δίνεται η δυνατότητα σε οργανώσεις παραγωγών να ε, εκτοπίσουν ενίσχυση εκκίνησης για κάθε τομέα πλην των οποροκυπευτικών. Γιατί πλην των απορροκυπευτικών, κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, διότι αυτά τα καλύπτει ο πρώτος πυλώνας για τα 12 κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πρόσφατα. Γιατί λοιπόν να μην διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής αυτής της τροπολογίας. Ε, για λόγους απλούστευσης και για λόγους διαφοροποίησης της μεταχείρισης, αλλά και για να μην επιβαρυνθεί με γραφειοκρατικό ε, φόρτο η εφαρμογή του κανονισμού. Έτσι λοιπόν προτείνουμε συγκεκριμένα να καλυφθούν όλοι οι τομείς για τα 27 κράτη-μέλη πλην του τομέα των απορροκυπευτικών. Θα μου επιτρέψετε να περάσω στον υπαριθμό 5 τροπολογία, τη λεγόμενη ευελιξία στο πλαίσιο της οργάνωσης κρατών περιφερειακού τύπου με στόχο την ε, αποφυγή απώλειας πιστώσεων. Το 2010, και ξέρετε ότι ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την ε, εξέταση των συνθήκων για αρκετά κράτη-μέλη, χορήγηση των πιστώσεων, αποδεικνύεται λοιπόν ότι η διαχείριση, η μεικτή διαχείριση, κοινή διαχείριση, μας επιτρέπει να αποφύγουμε αυτό τον κίνδυνο της αποδέσμευσης. Αφενός, αφετέρου, Πρόεδρε, η Επιτροπή επιμένει ώστε η αρχή διαχείρισης ενός προγράμματος να είναι εκείνη που θα έχει την ευθύνη και την πρωτοβουλία στην διαχείριση και τον έλεγχο. Και η ευελιξία που προτείνει η δική σας τροπολογία πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στην διάρρηξη αυτού του δεσμού μεταξύ αρχής διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσιονομικής. Εξού και η δική μας θέση, Πρόεδρε. Δεν θα ακολουθήσουμε δηλαδή τις δικές σας προτάσεις στην τροπολογία 5. Εν τέλει, όσον αφορά την τροπολογία τη σχετική με τον φόρο προσθέμενης αξίας, υπερθυμών 6, υπερθυμίζω ότι στις απαρχές αυτού του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια μεθοδολογία για τα διάφορα ταμεία. Δηλαδή, οι δημόσιες αρχές δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, ε, δεν θα μπορούσαν να έχουν ωφέλιμα ανάκτησης του ΦΠΑ. Γιατί. Διότι, αυτή ήταν η αρχική πρόταση όπως είπαμε, για όλα τα ταμεία. Σήμερα η κατάσταση αυτή ισχύει μόνο στο ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη αλλά και σε άλλα. Μερικά και βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει μεταβληθεί έτσι ώστε δεν μπορούμε να μιλούμε πλέον για ευθυγράμμιση. Οι, επιτροπές, οι υπηρεσίες λοιπόν της Επιτροπής αντιμετωπίζουν ε, το θέμα αυτό, μελετούν την υπόθεση ε, που μπορούμε να ακολουθήσουμε για την περίοδο μετά το 2013. Αυτό που κάνουμε είναι πάνω απ' όλα προσπαθούμε να ελέγχουμε το ποσοστό ε, εσφάλματος και τη διόρθωση που μπορούμε εμείς να επιφέρουμε στο δικό Αυτά πρόεδρε. Πανταζούμε, έχω καλύψει τις ε, τροπολογίες σας. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ιδιαίτερο χέρι η Επιτροπή για την σημειωμένη σύγκληση θέσεων μεταξύ ημών και ημών ε, στην πρόταση αυτή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι βουλευτές. E, Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά Σουσούβα. Φυσικά κατά εξαίρεση τροπολογιών ε, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις παρατηρήσεις. Αλλά εν συντομία, σε ό,τι αφορά την τροπολογία 3 για τα οπωροκυπευτικά, την είχαμε συμπεριλάβει διότι στο κείμενο υπάρχει ένα νέο στοιχείο, δηλαδή αναφέρεται ότι καμία στήριξη δεν θα ε, γιόμεθα στην Αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς εισάγετε. Ίσως εδώ να υπάρχει κάποια παρανόηση. Τώρα επίσης για το 5 καμία αλλαγή αλλά υπάρχει και το ζήτημα των κρατών μελών που επέλεξαν μια, μια περιφερειακή διαχείριση. Τότε η αποδέσμευση θα πρέπει να ισχύει. Ε, ευχαριστώ τον ε, κύριο Σουσούβα και αν δεν επιθυμεί κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο υπενθυμίζω πως ε, και εδώ η κατάθεση τροπολογιών Μάλλον προθυμεί η υπολογίων είναι 22 Μαρτίου στις 12 ε, το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Δεδομένου του ότι ο αντιπρόεδρος κ. Βαρσεμπόσκι θα καθυστερήσει, θα κάνουμε μια ελαφρά τροποποίηση της μισής διατάξεως. Αντί να περάσουμε στο σημείο 7, όπου η συγητής είναι ο αντιπρόεδρος ε, Βασεβόφσκι σχετικά με το ζήτημα του εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο μέχρι να φτάσει ο συνάδελφος. Το επόμενο σημείο είναι το σημείο 8. Επειδή βλέπω τον Λορέτσο Φωτάνα παρόντα, εάν συμφωνείτε θα κάνουμε αυτή την αλλαγή στην διάταξη. Περνάμε τώρα στο 8 και μετά θα επιστρέψουμε στο 7 για να μπορέσει το μεταξύ να έρθει ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Σημείο 8. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου σχετικά με βέβαια μέτρα ελευθέρωση για τα γεωτικά προϊόντα και τα προϊόντα αλίας. Εισηγητής ο συνάδελφος Λορέντσο Φοντάνα. Μόνο ότι η Επιτροπή διεθνού Εμπορίου είναι η αρμόδια τη ουσία Επιτροπή για θέματα εμπορικών συμφωνιών, το επενθυμίζω αυτό, η γνωμοδότηση τη Επιτροπής μα είναι ιδιαίτερη σημασία, διότι η συμφωνία με το Μαρόκο αφορά μια μεγαλύτερη απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών αγροτικών προϊόντων, μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, αλλά και προϊόντων αλίας. Η συνθήκη τη Λισαβόνα αύξησε σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και τώρα καλείται να δώσει την σύμφωνη γνώμη του στην σύναψη παρόμοιων συμφωνιών. Υπενθυμίζω πως από πλευράς ε, διαδικαστικής ε, θα πρέπει να κάνουμε σύσταση, να στείλουμε μάλλον σύσταση προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ως εκ τούτου απαιτείται τη στιγμή της ε, ψηφοφορίας να προκύψει μια ψήφος θετική η αρνητικη Μία απλή απόρριψη δεν θα επαρκούσε και θα σήμαινε ότι η Επιτροπή Γεωργίας δεν στέλνει καμία γνωμοδότηση στην Επιτροπή επειδή, μας έχει, επειδή έχει ζητηθεί από τον Επίτροπο Ντεγκούχτου, του προτείνω να αναβάλουμε την τελική ψηφοφορία αναμένοντας ε, την απάντηση του κ. Επιτρόπου. ω εκ τούτου, η προθεσμία κράτηση Ορπολογιών θα οριστεί συνάρτηση αυτού του γεγονότος. Τώρα να υπενθυμίσω σε σχέση με την ε, έκθεση του κ. Παπαστάμου που μεγκρίνει την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, παραμένουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με αυτές τις διμερείς συμφωνίες που συχνά θυσιάζουν ε, γεωργικά ζητήματα προς όφελος άλλων. Το έχουμε επανειλημμένο το, τονίσει και δεν θέλω τώρα να μιλήσω στη θέση του εισηγητή Φοντάνα και θα ήθελα να προτείνω εδώ ιδιαίτερη προσοχή. Εξάλλου έχει αναγγελθεί μια επιστολή του κυρίου Ατζής Καχνούκ, Υπουργού Γεωργίας του Μαρόκου και μόλις φτάσει η επιστολή θα την διανύμω στους συναδέλφους. Θα πρέπει να λάβουν λοιπόν υπόψη μια κατάσταση διάζουσα που διανύει το Μαρόκο, ομού με τις άλλες χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασρέκα σε αυτήν την κατάσταση της οικονομικοκοινωνικής κρίσης που έχει πλήξει την Αφρική. Αυτά είχα να πω, να δώσουμε αμέσω τον λόγο στον Λόριτζα Φοντάνα και μετά θα περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές και τους συνεργάτες που εργάστηκαν για τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης που υπενθυμίζω ότι θα περάσει στην Επιτροπή Ίντα και ε, ο συνάδελφος ε, Μποβέ σίγουρα θα μπορέσει να εμπλουτίσει τη συζήτηση που έχουμε και την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε μεταξύ μας. Θα ήθελα να συνοψίσω λοιπόν αυτά τα οποία προέκυψαν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, η πρόταση της Κομισιόν αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο βρίσκει το σύνολο των προσώπων με τα οποία συνομίλησα αντίθετο, διότι στον τομέα της γεωργίας κρίνουμε πως αυτά θα οδηγήσουν σε τεράστιες δυσκολίες για τις ε, γεωργικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για τις γεωργικές χώρες ε, της Μεσογείου, διότι θα δημιουργηθεί μια κατάσταση ανταγωνισμού που δύσκολα θα μπορέσουν να αντέξουν οι επιχειρήσεις μας και θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Να υπενθυμίσω πως ε, επανειλημμένα ετέθη το ερώτημα των ε, ε, φυτοφαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούν στις περιοχές αυτές της Αφρικής και που δεν χρησιμοποιούμε εμείς. Επίσης υπήρχε και ένα αίτημα το γεγονό ότι οι γεωργικέ ενδείξει δεν, δεν περιέχονται σε αυτήν την συμφωνία και έχουν ε, μεταρρυθεί για μερονικές συμφωνίες. Επίσης ε, υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες το ότι αυτή η πολιτική θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις ιδιαίτερα για περιοχές ε, οι γειτονικέ ε, του Μαρόκου και εδώ εξέφασαν ε, αντιρρήσεις ε, κάποιοι Ισπανοί συνάδελφοι αλλά και Ιταλοί αλλά και Έλληνες. Επίσης διάφορες οργανώσεις και είχα την ευκαιρία να δω ότι η Λάμπα Ζάιντα αλλά και άλλοι δήλωσαν ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι επιζήμια και για τους ε, γεωργούς του Μαρόκου. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις ε, συμφωνίες ε, διότι θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον κοινωνικές ε, δυσκολίες και εντάσεις ε, στις ε, χώρες αυτές, Μαρόκο κλπ. Άρα η γνωμοδότηση λοιπόν που θα στείλουμε στην Επιτροπή ίντα θα είναι μάλλον αρνητική, αλλά εν τόση θα θέλαμε να ακούσουμε αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ Λορέντσο. Έχει ζητήσει το λόγο ο Τζορτζ Λάιον και μετά Χέραντς Γκαρσία. Γιώργος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λορέντζο για τη δουλειά που έχει κάνει στην πρόταση αυτή. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό και σχετικά με τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας, όπου δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν θα τις καλύψουν ή όχι και θα τις συμπεριλάβουν στην Περιφερειακή Συμφωνία, ποτέ δεν μας έδωσαν απάντηση ξεκάθαρη. Και έτσι οι φιλελεύθεροι θα υποστηρίξουν την απόρριψη της πρότασης αυτής. Thank you. Ευχαριστώ, Τζορτζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Φοντάνα, για την άποψη που μας παρουσιάζει, δηλαδή να ζητήσουμε από την Εντροπή Διεθνούς Εμπορίου να καταψηφίσει την συμφωνία με το Μαρόκο. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά παράπονα σχέση με τη συμφωνία αυτά. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες όχι μόνο από τους παραγωγούς αλλά και από τον Όλαφ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα όπως το, η τιμή εισόδου. Υπάρχουν επίσης ε, και άλλες ανησυχίες από διάφορες επιτροπές, ε, κοινοβουλευτικές, ε, περιβαλλοντικά προβλήματα, προβλήματα υγείας κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να επιληθούν προτού να προχωρήσουμε. Για τον λόγο λοιπόν αυτό ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρόσβασή του και να πω ότι υπάρχουν αιτίε που αναφέρουν όχι μόνο η παραγωγή προκυφτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, πάρα πολλά προβλήματα που έχουν τεθεί. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να ε, σεβαστεί όλες αυτές τις θέσεις, ιδιαίτερα τις θέσεις των παραγωγών αλλά και των καναλωτών και να ε, ζητήσουμε να εφαρμόζονται τα διεθνή κριτήρια ποιότητας. Ευχαριστώ. Μάτω ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον ε, συνέλφο Φοντάνα για την ε, γνωμοδότησή του. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του κατά τη σύνταξη της ε, γνωμοδότησης. Να πω ότι κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι είμαστε κατά των συμφωνιών με τρίτες χώρες και με τις εμπορικές συμφωνίες στο σύνολό στού του τουλεχθέντος ε, είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε φυσικά να συμφωνήσουμε με συμφωνίες που πραγματικά είναι επιβλαβείς ε, και ζημιώνουν τα συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων Γεωργών και στην περίπτωση αυτή των Ισπανών Γεωργών. Αλλά και επηρεάζει πολλούς αγρότες των Καναρίων Ίσων, της Μούρτρια, της Ανδαλουσίας κλπ. Ω εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Επίση θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε κάθετοι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε τέτοιε συμφωνίε ενώ δεν τροποποιείται ο κανονισμό περί τιμών εισόδου, δεν ε, εγγυόμεθα. Μα εγγυάται μάλλον το βασίλειο του Μαρόκου την τήρηση κάποιων προποθέσεων και τέλο δεν ε, μας ε, εγγυώνται την αρχή της εμβαιότητας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αρχή της εμβαιότητας ε, που μόλι ψηφίσαμε στην Ολομέλεια με τις εκθέσεις Στάμπος Ο κύριος Δανέλη το λόγο και μετά τον Γκέλ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο να έχουμε μια μονοδιάστατη προσέγγιση στο θέμα αυτής της συμφωνίας. Απ' τη μια βεβαίως έχουμε την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία και το πλαίσιο που αυτή βάζει. Ε, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της αστάθειας της πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας της περιοχής αυτής. Ε, όμως παράλληλα έχουμε και ε, συγκεκριμένα προβλήματα στα οποία δεν έχουμε απάντηση. Έχουμε το πρόβλημα δηλαδή της διεθνούς νομιμότητας και αν αυτή τηρείται σε σχέση με την περιοχή της Σαχάρα. Ε, αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που συχνά συναντάμε σε παρόμοιες διμερείς συμφωνίες σε σχέση με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων γεωργικών προϊόντων. Εδώ είναι ένα μείζον ζήτημα, στο οποίο πολλές φορές έχουμε επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τις τα επίπεδα θα πρέπει να αναδιαμορφώσει τον τρόπο προσέγγισης των ε, διεθνών συμφωνιών, ε, διότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο γεωργικός τομέας να είναι ο μεγάλος χαμένος, ο μεγάλος ρηγμένος αυτών των συμφωνιών. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι μπροστά στα μείζωνα αυτά θέματα είναι εύκολο να πει ένα ναι ή ένα όχι. Ε, το περιθώριο που έχουμε μέχρι την ε, τελική έκφραση της ε, γνώμης μας θα μας, ίσως θα μας δώσει τη δυνατότητα με μεγαλύτερη, με μεγαλύτερη βεβαιότητα να αρνηθούμε την στήριξη ή να επισημάνουμε το ότι θα πρέπει εν τέλει να στηρίξουμε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να υπογραμμίσω όλε τι επιφυλάξει που ακούστηκαν για να πω ότι συμμεριζόμαστε και εμεί. Είπε βεβαίω ο Πρόεδρο ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δυσχερή μάλλον κατάσταση κυρίως ως προς τα κράτη της Μεσογείου, η κατάσταση μπορεί να μην ρυθμίζεται μέσα από αυτή την έκθεση, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι τις επιφυλάξεις αυτές και τους προβληματισμούς ε, με ακόμη περισσότερη πεποίθηση τους εκφράζω, καθώς βλέπω ότι είναι πολύ ενεργή η δράση των λόμπι και των ομάδων πιέσεως εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο. Εδώ, όσοι ασχολούμαστε με τα γεωργικά θέματα, πρέπει ή μη τι άλλο να εκφράζουμε τα θέματα που μας απασχολούν, τις θέσεις μας, τα συμφέροντα που θέλουμε να προαγάγουμε και να μην αφήνουμε πιέσεις θέλει να μας υποχρεώνουν ε, σε σύναψη συμφωνιών οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον της γεωργίας. Η συζήτηση στην ε, ολομέλεια στο Στρασβούργο που είχε να κάνει με τη συμφωνία τη σχετική με την Κορέα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, την παρακολούθησε από την αρχή μέχρι το τέλο και ο Επίτροπο Φανγκιούχτ δεν ε, χρησιμοποιήσετε μία λέξη για τη Γεωργία, ούτε καν τον όρο Γεωργία δεν άκουσα από τα χείλη του. Μόνο βιομηχανικά προϊόντα, υπηρεσίε ήταν αντικείμενο τη συζήτηση. Από την άλλη, βέβαια, κάθε συμφωνία έχει επιπτώσεις και για τη γεωργία μας για τη γεωργική πολιτική. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε επαρκώς υπόψη. Δεν θέλω λοιπόν να πω τίποτε περισσότερο αυτή τη στιγμή, ίσως να χρειαστεί να απορρίψουμε, ίσως να αποφασίσουμε να υποστηρίξουμε, αλλά πάντως θα πρέπει να είμαστε θέση να κοιτάξουμε όλες τις συνθήκες και να τις εκτιμήσουμε συνολικά. Είμαι τώρα προς το παρόν διατεθειμένη να συζητήσω, να διαπραγματευθώ, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια ευκαιρία να προχωρήσουμε κατά τρόπο ευκταίο. Διαφορετικά θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση. Ζωζέ Μποβέ και μετά Ρουίς Καπουλεσάντος. Μποβέ. Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας λαμβάνω το λόγο και τι είμαι εισηγητής της Επιτροπής για το Εθνές Εμπόριο στην υπόθεση αυτή. Με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολουθώ τα όσα λέγονται. Ιδιαίτερος εκτιμώ τις προτάσεις του κυρίου Φοντάνα, μου φαίνονται ισορροπημένες, σωστά και ότι κάποια σημεία ίσως χρειάζονται περισσότερη προβολή. Φερρυπίν, δομή του εξωτερικού εμπορίου. Όλοι γνωρίζουμε, όπως οι συνάδελφοι της Επιτροπής, ότι όποιος εξάγει σήμερα και Φερρυπίν. Από το Μαρόκο προς την Ευρώπη έχουμε να κάνουμε με εξαγωγές μεγάλων δομών. Αυτός που εξάγει λοιπόν προς την Ευρώπη δεν είναι ένας μικρός παραγωγός, είναι μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Και έχουμε εδώ Φερρυπίν στην περίπτωση του Μαρόκου με μια, να κάνουμε μια μεγάλη επιχείρηση που είμαστε Αζούρα. Επιχείρηση που όχι μόνο έχει συμμετοχή και ευρωπαϊκών κεφαλαίων, για το οποίο δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά, και εδώ ακριβώς είναι το κύριο πρόβλημα, εδρεύει στη Δυτική Σαχάρα. Σε εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Εδώ ακριβώς έχουμε το ζήτημα ουσίας και γι' αυτό και το ζήτημα των εξαγωγών μέσα από το, από το, νομικό πλαίσιο του Εθνούς δικαίου είναι ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Και όταν έθεσα το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπολίου για να ζητήσω να παρακολουθήσουν πρώτα η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου αλλά και αντίστοιχα οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα αυτό για να δούμε αν υπάρχει όντω νομικό ζήτημα προ το διεθνέ εμπόριο ποια είναι η θέση του Μαρόκου, τι είναι το Μαρόκο, μέχρι πού, ε, πού τελειώνει η επικράτειά του, πού αρχίζει. Όμω φαίνεται ότι ο κύριο Δεγκούχτ, ο επίτροπο για το Εξωτερικό Εμπόριο, δεν είναι εις θέση σήμερα να μα πει ποια είναι η απάντηση. Μα λέει δεν είμαι αρμόδιο η κυρία Άστον θα πρέπει να απαντήσει. Και αν δεν είναι η κυρία Άστον αρμόδια, ποιο θα έρθει να δώσει απάντηση εν τέλει. Η κατάσταση είναι ε, γελία θα έλεγα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιλύσει το πρόβλημα. Ο Ρόμπερτ ε, υπουργό για το εξωτερικό εμπόριο, πριν από χρόνια τον γινόταν η συζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Μαρόκου με τις διαπραγματεύσεις, έλυσε το πρόβλημα μια ξεκάθαρη ε, διαχωριστική γραμμή. Εμεί λοιπόν πολιτική συζήτηση στην, ε, πολιτική τοποθέτηση μάλλον στη συζήτηση αυτή θα λάβουμε. Είναι ένα άλλο αντικείμενο. Αλλά για το εξωτερικό εμπόριο πρέπει να μην παραβλέψουμε ορισμένα πράγματα τα οποία επιπλέον δυσκολεύουν καθώς εάν μα δοθεί η απάντηση ότι δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικέ γραμμέ τότε ούτε η πρώτη εμπορική συμφωνία είναι σαφής. Άρα έχουμε ένα συνολικό πρόβλημα συμφωνιών εμπορικών με το Μαρόκο. Αυτέ τι ολίγε παρατηρήστε θέλω να ε, διατυπώσω. Σήμερα δεν ξέρουμε πότε θα λάβουμε απάντηση στο θέμα αυτό. Σε 15 μέρε, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Πρωταρχικό ερώτημα, πρόκριμα από πλευρά του Κοινοβουλίου, ήταν ένα ερώτημα το οποίο ε, στο οποίο δόθηκε απάντηση τρει μήνε μετά, γιατί ήταν περίπλοκο. Αυτά ήθελα να σα δώσω σαν πληροφορίε, τελευταίε εξελίξει, για να επισημάνω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, διότι έχουμε να κάνουμε και με το μέλλον του μικρού παραγωγού του Μαρόκου ή τη Τινησία της τη Αιγύπτου, τελευταία ανάλυση, και με θέμα κεντρική σημασία. Έχουμε να κάνουμε μια συμφωνία στην οποία παρότι έχουμε ήδη συζητήσει με οργανώσει παραγωγών του Μαρόκου που είχα την ευκαιρία να δείσω στο Στρασβούργο, ε, δεν βλέπω δυστυχώ να αποβαίνει αυτή η συμφωνία όφελό του. Ακριβώς αυτό σκέφτεται και ο Υπουργός του Μαρόκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι εύκολο να παίρνει κανείς το λόγο, να μιλάει, να σχολιάζει. Εφόσον θέλουμε απλά να λειτουργούμε σαν συνδικαλιστές του γεωργικού τομέα της Ευρώπης. Δεν είναι όμως αυτή η δουλειά μας, θα πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο το βόρειο τμήμα της Αφρικής καίγεται. Έχουμε εμείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τις χώρες αυτές και ιδιαίτερα με το βασίλειο του Μαρόκου, το οποίο μέχρι τώρα σαν καθεστώς έδειξε μια κάποια μετριοπάθεια θα έλεγα και ένα σχετικό πολιτικό άνοιγμα σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλα καθεστώτα της περιοχής. Το να απορρίψουμε λοιπόν απλά την πρόταση αυτή όπως προτείνεται από τον εισήγητη μου φαίνεται μια, μια λύση η οποία είναι λανθασμένη και δεν ε, εξυπηρετεί ε, ούτε τους στόχους της Επιτροπής μας. Προφανώς και θα πρέπει να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις που να λαμβάνουν υπόψη και τα πιο ευαίσθητα προβλήματα. Αλλά το να διακόψουμε κάποιες εμπορικές σχέσεις οι οποίες λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βοηθάει η συμφωνία αυτή επαγγελματικά τους Μαροκινούς, νομίζω ότι είναι προβληματικό. Νομίζω ότι όλοι θα φυγούν και οι μικροί εξαγωγείς και συνολικότερα ο τομέας. Ο τομέας ο γεωργικός ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για το Μαρόκο, ακριβώς γιατί απασχολεί ένα τεράστιο αριθμό εργαζομένων, εργατικού δυναμικού. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει τα πράγματα να τα δούμε και λίγο διαφορετικά. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνατόν έτσι ώστε η συμφωνία να υπάρξει, να λειτουργήσει, αλλά με ισορροπημένο τρόπο, με τρόπο ο οποίος να σέβεται τους κανόνες στον τομέα της υγείας κτλ. Και θα ήταν σοβαρό λάθος εμείς να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή. Πράγματι δύσκολη θέση μας. Ταραμπέλα κάποια επιπλέον στοιχεία ακριβώς στα πλαίσια αυτών που είπε και ο Λουίς. Να σας θυμίσω ότι το 86 όταν μπήκε η Ισπανία και η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά φορτοϊγά ισπανικά και πορτογαλικά τα απαγόρευαν να μπουν στη Γαλλία οι Γάλλοι παραγωγή ε, που φοβόντουσαν τη γεωργική παραγωγή. Λοιπόν, θα πρέπει να μπούμε στην θέση αυτών που είναι ε, διστακτικοί σε σχέση με μια τέτοια συμφωνία με το βασίλειο του Μαρόκου. Να επιστήσω την προσοχή σας όμως ότι στα πλαίσια όλων των συμφωνιών που μπορούμε να υπογράψουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ότι η νότια πλευρά της Μεσογειακής Λεκάνης πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα όχι μόνο λόγω εγκύτητας, αλλά είναι θα έλεγα προτιμησιακές οι σχέσεις που έχουμε με αυτή την περιοχή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ταχθούμε στη συμφωνία αυτή, θα πρέπει να κάνουμε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον κανονισμό για τις τιμές εισόδου, γιατί έχει γίνει ουσιαστικά ταμπού σε σχέση με ε, ε, τα, με το βόλιο κρέας και με την παραγωγή οποροκυπευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ένωσης. Σχετικά τώρα με τη Δυτική Σαχάρα, λίγα λόγια. Κάθε φορά που μιλάμε με το Μαρόκο επανέρχεται το θέμα. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε μία στάση σε σχέση με την παραγωγή προϊόντων και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί θα έχουμε να εξετάσουμε και τη Συμφωνία της Κολομβίας, οπότε και αυτά θα τεθούν εκ νέου. Τώρα λέω η Κολομβία, θα μπορούσα να μιλήσω και για άλλες χώρες. Γιατί ξέρετε ότι εκεί συνεχίζουν να δολοφονούν αυτούς του συνδικαλιστές που υπερασπίζονται τους εργαζόμενους και στον τομέα της γεωργίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να τροπολογηθεί η συμφωνία αυτή και δεν θα πρέπει να απορριφθεί έτσι μιάς γιατί οι εταίροι μας στην νότια πλευρά της Μεσογειακής κάνεις θα ερμηνεύσουν την κίνηση αυτή σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός των κοινωνικών κανόνων κτλ. Διερωτώ με αν οι Πακιστανοί οι οποίοι δουλεύουν στη Φλάνδρα ή οι Μαροκινοί οι οποίοι δουλεύουν στην Ισπανία και στην Ανδαλουσία έχουν κοινωνικά επίπεδα προστασίας ευρωπαϊκού επίπεδου και ε, κατοικίες οι οποίες ε, να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτό και δεν το κάνουμε συνήθως. Ευχαριστώ Μάρκ. Θα δώσω το λόγο στον Κουτιέβες. Η δυσκολία Μάρκ είναι αυτή. Εμείς δεν μπορούμε να τροπολογήσουμε. Αυτό είναι το δράμα ναι. της κατάστασης. Πρέπει να πούμε μόνο ναι ή όχι. Η δυσκολία λοιπόν αυτή είναι. Πρέπει να φανούμε συνεκτικοί ή θα πρέπει να φανούμε ευαίσθητοι. Δεν έχουμε περιθώρια διαφοροποίησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους και ιδιαίτερα με τον σοσιαλιστή συντονιστή. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα να, ως Επιτροπή Γεωργίας να αναρωτηθούμε αν αυτή η συμφωνία είναι χειρότερη από αυτήν που υπογράψαμε το 2003 και δεύτερον τι θα συμβεί με τον κανονισμό 2003 εάν αυτός ο κανονισμός απορριφθεί από το Κοινοβούλιο εάν θα επανέλθουμε σε αυτήν τη συμφωνία του 2003 δηλαδή Κρίνω λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία βελτίωσε σημαντικά την συμφωνία που είχαμε υπογράψει με το 2003. Τις ποσοστώσεις, τιμές ε, εισόδου, ρήτρα προφύλαξης ε, κάθε συμφωνία μπορεί να προκαλεί ορισμένες ανησυχίες ε, σε κάποιους κλάδους. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτός ο κλάδος ε, απελευθερώνει τα ευρωπαϊκά προϊόντα που πολλούνται στο Μαρόκο κατά ένα σημαντικότερο ποσοστό. Τώρα, αν ακούσουμε τις ανησυχίες ε, αναφορικά με τις ποσοστώσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ντομάτα. Να υπενθυμίζω ότι αυτή η αύξηση αφορά μόνο το 0,6% της ευρωπαϊκής ποσότητας. Μιλώντας για τους ελέγχους της τιμές εισόδου, υπενθυμίζω ότι οι έλεγχοι των τιμών εισόδου εμφαίνονται στην προνόμενη συμφωνία και υπάρχει και μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού των τιμών εισόδου του Συμβουλίου μεταξύ Αυτόν ε, περιλαμβάνεται και η Ισπανία. Πρέπει να είμαστε λοιπόν κάπως σοβαροί και αυστηροί όταν ε, μιλάμε για πολιτικά θέματα. Τώρα, ο έλεγχος της συμφωνίας ε, και μας και ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι η προηγούμενη συμφωνία δεν εφαρμόστηκε πλήρως. Γι' αυτό πρέπει να απορρίψουμε και αυτήν. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να έχουμε στόχο την ε, προσπάθεια εποπτείας ε, και ελέγχου της εφαρμογής των κανονισμών. Ειδικά για μια συμφωνία όπως αυτή που είναι τόσο σημαντική 7. Νομίζω ολοκληρώνουμε εδώ με την Μαρία Μεγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τις λεπτομέρειες συμφωνίες αυτές θα στηριχθώ βέβαια στι ε, ειδικέ γνώσει που έχουν να συνάδελφοι από την, ε, τις που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Αλλά γενικότερα για τη συμφωνία θα ήθελα να ρωτήσω εάν θέματα της γεωργίας Πιστεύετε ότι δεν δόθηκε αρκετή προσοχή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι συνέπειε που μπορεί να έχουν οι εμπορικέ συμφωνίε εν γέννη στον τομέα τη γεωργία και ιδιαίτερα όσον αφορά τι προδιαγραφέ παραγωγή, ε, την ε, χρήση των εισαγωγών αυτών και τις επιπτώσεις του στα λεγόμενα μη εμπορικά ζητήματα. Και βέβαια εδώ θα βάλω και το θέμα της ευημερία των ζώων. Σημειώνω επίσης ότι οι συνάδελφοι ιδιαίτερη ανησυχία έχουν εκφράσει για τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία και συμμερίζομαι την ανησυχία. Ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να αποφασίσουμε αν θα πούμε το ναι ή το όχι. Δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε εδώ πέρα τη συμφωνία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση ασφαλώς. Ε, θα υπενθυμίσω όμω την κατάσταση που έχουμε να κάνουμε και με το βόλιο κρέα, αγωγέ βόλιο κρέατος από την Βραζιλία. Πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε συμφωνία εμπορική. Είχαμε, είχε δοθεί άδεια για εισαγωγή βοήου κρέατο από τη Βραζιλία και χρειάστηκε με πολλέ προσπάθειε και χρόνο βέβαια που δαπανίσαμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έπρεπε να απαγορεύσει τι εισαγωγέ βοήου κρέατο από τη Βραζιλία. Άρα Ξέρω ότι δεν είναι ο δρόμος ανοιχτός, δεν είναι τα πράγματα ε, δεν προχωρούν απρόσκοπτο όλα αυτά. Πρέπει να κάνουμε αγώνα και να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αντιληφθεί τι ανησυχίε μα. Και δεν έχω πιστεί ότι η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τι ανησυχίε μα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσει τι λεπτομέρειε τη την έκθεσή μα η Επιτροπή, την έκθεση τη προηγούμενη εβδομάδα και να λάβει υπόψη τι ανησυχίε τη δικέ μα, του γεωργικού τομέα ευρύτερα. Επίση, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το συμφέρον του παραγωγού, αλλά και του καταναλωτή, του εργαζομένου. Έχει να κάνει με τα, με τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη και δεν νομίζω ότι μπορούμε να προάγουμε την ιδέα του εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών πάση θυσία και με κάθε τίμημα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν... δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς έχουμε εγκρίνει την έκθεση Παπαστάμκου και μάλιστα με ευρυτά τη συμμετοχή και στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ήταν μια πολύ σημαντική έκθεση της αμοιβαιότητα των νόμων, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση έχει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν μιλάμε για το Μερκοσούρι, για την Ασία, μιλάμε για το Μαρόκο, και στα πλαίσια της δύσκολης κατάστασης που ζει αυτή η περιοχή προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε με κανένα τρόπο να μην συνεισφέρουμε στη χειροτέρευση της κατάστασης. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε επίσης ότι σε επίπεδο διμερών συμφωνιών εμείς είμαστε υπέρ των πολυμερών βέβαια συνδέσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο διμερές, ειδικά για τη γεωργία, τα προβλήματα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολλά. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο κύριε Φοντάνα, ας μην καθορίσουμε την ημερομηνία για τις τροπολογίες αν δεν έχουμε μια διαφορετική απάντηση από την Επιτροπή. Πριν δώσω πάλι το λόγο στο Λορόνσο, ζητώ από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κλάρκ, αν θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των μελών της Επιτροπής σας, να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Και ίσως να προσπαθήσω να διορθώσω κάποιες, ε, ε, κάποιες ανακρίβειες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη συζήτηση αυτή. Αρκετοί συνάδελφοί σας αναφέρθηκαν στο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο αναγκαστικά κινούμεθα σε μια περιοχή η οποία βιώνει μια σημαντική κρίση και όπου το Μαρόκο εξακολουθεί να είναι θα έλεγα φάρος ε, ασφαλής για την περιοχή ακόμα και σήμερα και με αρκετές σημαντικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις και το Συμβούλιο μάλιστα καλωσόρισε τον οδικό χάρτη τον οποίο ακολουθεί το Βασίλειο του Μαρόκου στην τελευταία του συνεδρίαση. Λοιπόν, σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, όπως είπαν και ορισμένοι συναδελφοί σας, πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ επιφυλακτικά σε σχέση με το μήνυμα που θα στείλουμε στο Μαρόκο σαν χώρα εταίρος στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Θέλουμε σαν Επιτροπή να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή. Θέλουμε να υπάρξουν περισσότεροι μετανάστες από το Μαρόκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να υπάρξουν λιγότερα ή περισσότερα γεωργικά προϊόντα. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε από όλα αυτά ή τι δεν θα πετύχουμε αν απορρίψουμε τη συμφωνία. Για την Δυτική Σαχάρα Συμφωνώ με τον Ζωζέ Μποβέ και όσους άλλους είπαν ότι εμείς, εσείς και εμείς, ε, εσείς μάλλον αξίζετε μια πιο ξεκάθαρη άποψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ να δώσω μια τέτοια απάντηση αυτή τη στιγμή αμυνόμενος θα έλεγα. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με τη συμφωνία αυτή και με το τι ισχύει ακριβώς με την προηγούμενη συμφωνία σχετικά με την Δυτική Σαχάρα. Μια ξεκάθαρη απάντηση ελπίζω να σας δοθεί σε λίγες ημέρες και ελπίζω να δούμε και τι συνέπειες μπορεί να προκληθούν από την απάντηση αυτή. Αν πράγματι καλύπτεται de facto η Δυτική Σαχάρα από την εμβέλεια της συμφωνίας ή όχι. Λοιπόν, περιμένετε κι εσείς την δική μας απάντηση πριν επισημοποιήσετε την τελική σας θέση. Συγγνώμη που καθυστερώ λίγο, αλλά ίσως να προσπαθήσω να διορθώσω και ορισμένες παρανοήσεις σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Καταρχάς, στην γνωμοδότηση, στην αρχή της γνωμοδότησης λέγεται ότι η συμφωνία αυτή είναι ασημετρικού χαρακτήρα υπέρ του βασιλείου του Μαρόκου. ότι το Μαρόκο πρέπει να ε, φιλελευθερωποιήσει το 45% των εισαγωγών του και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 55%. Αυτό είναι αλήθεια σε αριθμητικό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργήσει η συμφωνία πλήρως. Εμείς θα παραμείνουμε στο 55% των προϊόντων από το Μαρόκο, αλλά το Μαρόκο θα πρέπει να φτάσει στο 70% ε, των ε, εισαγωγών απελευθερωμένων από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Να λοιπόν, που βρίσκεται η, περί, που βρίσκεται η πραγματική ασυμμετρία. Είναι σαφέστατα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες αναφορές σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής στην πολιτική ανταγωνισμού και στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Όταν κάποιος εξετάσει τη συμφωνία και την αύξηση των εισαγωγών σε βασικούς τομείς, σε σχέση με το σύνολο της ευρωπαϊκής παραγωγής, νομίζω ότι τα πράγματα παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο. Αν εισαγωγή σκόρδου θα αυξηθεί η εισαγωγή κατά 0,25%. 1,6% η εισαγωγή αγκουριών, 6% η εισαγωγή ε, σε ντομάτες, ε, κολοκυθάκια 1, κάτι πάλι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο απειλεί την γεωργική ε, βιομηχανία και τη γεωργική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, έγιναν ορισμένες αναφορές ε, στα κοινωνικά επίπεδα και στο μη σεβασμό από πλευράς του Μαρόκου ε, των κανόνων παραγωγής στον τομέα της υγείας και υγιεινής. Ε, πρώτον, όπως και στα πλαίσια κάθε διεθνούς συμφωνίας, το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των καταναλωτών δεν θα επηρεαστεί σε καμία περίπτωση. Οι κανόνες μας θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως. Δεν υπάρχει καμία ειδική ρύθμιση και υποχώρηση προς το Μαρόκο. Το Μαρόκο καλείται να σεβαστεί ε, τις ισχύουσες ε, ε, συνθήκες παραγωγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, έχουμε κάνει κάποιες μελέτες επιτόπου στο Μαρόκο και είδαμε ποιο είναι το επίπεδο ζυζανιοκτώνων τα οποία χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που εξάγει το Μαρόκο και υπήρξαν ορισμένες προειδοποιήσεις και είδαμε ότι τα τρία τελευταία χρόνια 19 μόνον φορές υπήρξε ένα σύστημα, το σύστημα κινητοποίησης, ενώ το σύστημα αυτό κινητοποιήθηκε 30 φορές για την Ισπανία. Πριν λοιπόν ασκήσουμε κριτική στο Μαρόκο για μη σεβασμό και τήρηση των κανόνων SPS στον τομέα της υγείας και υγιεινής θα πρέπει να κάνουμε τις απαιτούμενες προσαρμογές στο εσωτερικό μας. Τελευταίο σημείο, Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή είναι θα έλεγα ιδιαίτερα μικρή σε επίπεδο. Θα αυξηθεί το επίπεδο προς η παραγωγή της ντομάτας στην Ευρώπη κατά 50.000 τόνους. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια παραγωγή η οποία δεν θα απειλήσει καθόλου την ευρωπαϊκή γεωργία Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό και θα το ξαναπώ στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Παρακαλώ να βλέπετε τα πραγματικά στοιχεία και ίσως να καταλήξετε κάποια από εσά σε διαφορετικές απόψεις από αυτές τις οποίες παρουσιάσατε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Κλάρκ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Φοντάνα για να κλείσει παρακαλώ και μετά θα επανέλθουμε στο 7 γιατί ο Αντιπρόεδρος Βασιεβόσκη είναι μαζί μας. Καταλάβαμε ότι η Ισπανία είναι πιο επικίνδυνη από το Μαρόκο. Λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα. Ίσως να έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση. Εμείς ε, πρέπει να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συμφωνία, αλλά μακριά από μένα κάτι τέτοιο σε ό,τι πάλι συμφωνία με το Μαρόκο. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένο θέμα και επειδή δεν μπορούμε να πούμε μόνο ναι ή όχι και παρατηρώντας το ενδιαφέρον που έχουμε ως Επιτροπή Γεωργίας, άποψή μου είναι ότι η γνωμοδότησή μας ε, δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να βελτιώσουμε την συμφωνία, αλλά εμείς ε, σε αυτό το επίπεδο και με αυτή την γνωμοδότηση δεν μπορούμε να το πράξουμε. Χρειάζεται λοιπόν ε, επί της να στείλουμε, μάλλον στείλουμε μια γνωμοδότηση, επί της ουσίας είναι αρμόδια η Επιτροπή ίντε και ο κ. Μποβέ να πούμε ότι η γνωμοδότηση αφορά την θέση μας ως ε, Επιτροπή και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ θα αξιολογηθεί. Αλλά δεν μιλάμε για το σύνολο της Συμφωνίας του Μαρόκο. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Διαφορετικά αυτή θα ήταν ε, και η πρώτη στη προσπάθειά μου, το πρώτο στο μέλημά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λορέντσο. Μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο 7 τροποποίηση της οδηγίας 297 ε, για την ε, κατανοϊκό πυρετό των προβάτων ε, Γιάννους Καταμπόφσκι είναι εισηγητής να πω πρώτα ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κατεπήγον λόγω της επικείμενης περίοδου εμβολιασμού που θα ξεκινήσει τον Μάιο. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετηθεί στις 4 Απριλίου η εκθεσή μα στο Στρασβούργο. Γι' αυτό ζήτησα να τεθεί στη μέσα διάταξη τη Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της λόγω εβδομάδος. Έτσι θα οριστικοποιήσουμε το θέμα κατά τη διάρκεια τη Ολομέλειας του Μαΐου. Τώρα εδώ υπάρχει το θέμα των ε, πινάκων αντιστοιχίας correlation table που προτείνονται από την Κομισιόν αλλά τις αρνείται το Συμβούλιο. Τις απέριψε να επενδυμίσω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να τονίσει τη σημαντική συμπερίληψη αυτών των ε, πινάκων ε, ανησυχία στην οδηγία. Αυτή η θέση βιώθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στην συνάντηση τη 25η Νοεμβρίου 2010 και ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο και την Κομισιόν σε μια επιστολή που υπόγραψε ο πρόεδρο Μπιούζεκ στι 9 Δεκεμβρίου. Θεωρώ λοιπόν πω η Επιτροπή μα θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτή τη θέση γιατί είναι ευθύς αμέσω τον λόγο αντιπρόεδρο κ. Βοζεμπόφσκι. Γιάννο, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επισημάνατε ίδια εσείς τα κύρια προβλήματα που είχα να αντιμετωπίσω στην έκθεσή μου σε σχέση με την οδηγία αυτή. Είναι ξεκάθαρα νομίζω τα δεδομένα. Έχουμε να κάνουμε με την τροποποίηση της οδηγίας έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα νέα και καλύτερα ε, εμβόλια ε, για το καταρροϊκό πυρετό, κυρίως στην Νότια Ευρώπη όπου έχει μεγαλύτερη διάδοση η νόσος. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω συζητήσει και ε, κάτι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσω να εξασφαλίσω ότι η επιταχυμένη αυτή διαδικασία μέσα στο Κοινοβούλιο θα ε, γίνει ε, χωρίς προβλήματα και συνέπειες ότι δεν υποκρύπτεται τίποτε δηλαδή πίσω από την επιτυχημένη διαδικασία. Οι όποιες επιφυλάξεις μου έχουν διασκεδαστεί εντωμεταξύ και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε την προσαρμογή της οδηγίας για την καλύτερη για τον καλύτερο εμβολιασμό των ζώων στην Νότια ε, Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Εάν μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη ανάγνωση μέσα στην ε, Ολομέλεια του Απριλίου, τότε θα μπορέσει εγκαίρως και πριν από την φερινή περίοδο ε, του 2011 να γίνει ο εμβολιασμός. Άρα θα έχουμε κερδίσει ένα χρόνο. Δεν Θα χρειαστεί να πέρασει ένα ολόκληρο χρόνο για να γίνει ο εμβολιασμό. Όπω είπα, όμω υπήρχε ένα πρόβλημα ω προ τον πυρήνα των αντιστοιχειών Πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη οδηγία. Υπάρχει γενικά ένα ζήτημα των πρακτικών που ακολουθούνται και πολύ σωστά επεσήμανε ο Πρόεδρος ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του μέσα από μια επιστολή του Πρόεδρου Μπούζεκ που έχει εγκριθεί και από τη διάσκεψη των Προέδρων στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι σε κάθε οδηγία θα πρέπει να, προσα... να προ επισυνάπτεται ένας πίνακας ε, αντιστοιχειών των ε, νομοθετημάτων τα οποία ε, υιοθετήθηκαν προκειμένου να ε, ενταχθεί η συγκεκριμένη οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Έχει λοιπόν δεχθεί το Κοινοβούλιο αυταίου στους πίνακες της έχει προσαρμόσει τις εργασίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε, ως εκ τούτου θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα προηγούμενο που θα πρέπει να ακολουθείτε από εδώ και μπρος. Θέλουμε δηλαδή η οδηγία αυτή να έχει και πίνακα αντιστοιχειών. Είχα σήμερα την ευκαιρία να εξετάσω τις τελευταίες εξετάσεις, εξελίξεις, συνεργασία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να πω ότι από πλευράς του Συμβουλίου εκφράζονται ορισμένες ανησυχίες ως προς τους πίνακες αντιστοιχίας και ότι σκοπεύει το Συμβούλιο να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Πάντως εγώ ως ε, υποστηρίζω αυτή την ιδέα των πινάκων αντιστοιχίας διότι πρόκειται για μέτρο το οποίο θα βελτιώσει τη διαφάνεια ε, και θα επιτρέψει να επαληθεύσουμε σε κάθε περίπτωση εάν το ε, εθνικό δίκαιο έχει σωστά προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό. Γιατί συχνά ε, παραγνωρίζονται κάποιοι κανόνες και θα πρέπει πάντα να είμαστε θέση να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ή μεταφράζεται στο εθνικό δίκαιο μια ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα με τον πίνακα αυτό, τον πίνακα της ίδιας διαθεσή μας, θα μπορούμε πολύ εύκολα να διαπιστώσουμε ε, εάν έχει γίνει σωστή ε, εφαρμογή. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι εάν το Σύμβουλο δεν δεχθεί αυτή την ιδέα του πίνακα αντιστοιχίας, θα έχουμε πρόβλημα, θα χρειαστεί να περάσουμε σε ε, τρίτη ανάγνωση και άρα θα καθυστερήσει αυτή η οδηγία να μπει σε εφαρμογή. Θα περάσουμε το Μάιο και θα έχουμε χάσει τη συγκεκριμένη περίοδο εμβολιασμού, τη φετινή δηλαδή. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι συμφωνώ με τις θέσεις του Προέδρου. Δεν θα πρέπει το θέμα αυτό να ε, προσκρούσε στο μόνο ζήτημα του πίνακα αντιστοιχειών. Θα ήταν καλό φυσικά να τους έχουμε. Ας δούμε γενικά ποια είναι η κατάσταση και ποια ε, θέση θα εκφράσει το Συμβούλιο, ενδεχομένω και να συμφωνήσει εν τέλει μαζί μα, ώστε να μπορέσει να τεθεί το ταχύτερο δυνατό χωρίς προβλήματα η οδηγία. Ευχαριστώ κύριε Βατσεβόσκη. Λίζαμπετ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ του ΕΛΚΑ Θέλω να επισημάνω ότι πρώτα απ' όλα οφείλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, έκανε πολύ καλή δουλειά. Τίποτε το ουσιαστικό δεν έχουμε να τροποποιήσουμε στις προτάσεις του ή να αντιτάξουμε, τον υποστηρίζουμε λοιπόν. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω κάτι το οποίο κατέστησε σαφές το, ε, τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις τώρα. ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε αυτό ενθαρρύνω τον ε, εισηγητή μας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή τη λύση της ε, του πίνακα αντιστοιχειών, γιατί είτε πρόκειται για την Επιτροπή, είτε για το Συμβούλιο, είτε για μας έχουμε όλοι μας ευθύνη στην ουσιαστική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Και γι' αυτό ρωτώ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι δυνατόν ε, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ο καθένας μας από πλευράς του. Δεν πρέπει να συζητήσουμε όλοι με όλους και να ακούσουμε όλοι τα επιχειρήματα των ε, λοιπόν. Σε αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή που έκανε τη σχετική προσπάθεια. Γιατί πραγματικά βλέπω να κάνει ό,τι μπορεί έτσι να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Που είναι βέβαια δύσκολο θέμα, το θέμα της εφαρμογής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την προσπάθεια, για την προσπάθεια την οποία έκανε ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι αναζητεί μια κάποια συμφωνία και προσπαθεί να απομακρύνει τις δυσκολίες που υπάρχουν. Να υπογραμμίσω εδώ δύο θέματα. Ακόμα και αν πρόκειται για μια έκθεση η οποία δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην Επιτροπή μας, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι έχει μεγάλη σημασία για τον τομέα της εκτροφής ζώων, γιατί το νέο αυτό εμβόλιο που είναι στόχος τροποποίησης της οδηγίας επιτρέπει πράγματι από ό,τι φαίνεται να προλάβουμε και να ξεπεράσουμε κάποιες επιδημικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κοντά στην Αφρική και να αποφύγουμε έτσι και μία κυκλοφορία του συγκεκριμένου ιού, διευκολύνοντας τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί στις συγκεκριμένες ζώνες, ζώνες με περιορισμούς κτλ. Ο Αντιπρόεδρος το έλεγε πολύ σωστά αυτό και συμμερίζομαι με την άποψή του για τους πίνακες αντιστοίχησης Νομίζω ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να διευκολύνει την διαδικασία σύνταξης αυτών των πινάκων. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μία βελτίωση, το κείμενο είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, το εμβόλιο είναι, το αδρανές αυτό εμβόλιο είναι επίσης καλύτερο από ό,τι υπήρχε διαθέσιμο, θα πρέπει πριν το καλοκαίρι να τεθούν σε εφαρμογή και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι οι πίνακες αντιστοίχησης να μην θέσουν εμπόδια και οδηγήσουν στην καθυστέρηση της διαδικασίας και εμβολιασμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αργά για να μπορέσετε να φορέσετε τα ακουστικά σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο για μια εξαιρετική προσπάθεια την οποία έκανε. Να μην ξεχνάμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα ζώα και για τους γεωργούς ο εμβολιασμός να γίνει φέτος. Δεν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά αποκλειστικά τον νότο της Ευρώπης. Θυμίζω ότι μετά από δύο ζεστούς χειμώνες, τους οποίους ζήσαμε, στις αρχές αυτής της δεκαετίας αντίστοιχες εκδηλώσεις α, καταρροϊκού πυρετού είχαμε και στη Σουηδία. Είναι μια ασθένεια η οποία διαδίδεται στο σύνολο της Ευρώπης, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε και να το φανταστούμε πριν δέκα χρόνια. Ας χρησιμοποιήσουμε την διαθέσιμη τεχνολογία λοιπόν, για να εκριζώσουμε επιτέλους την ασθένεια αυτή και να εμποδίσουμε ε, να υποφέρουν τα ζώα και οι άνθρωποι. Ευχαριστώ κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εδώ στο καταλογικό που υπηρετώ είμαστε στην πρωτοπορία του αγώνα ώστε να αποτρέψουμε την είσοδο της ζωνός στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντοτε ακούγονταν επιφυλάξει για το αν αυτή η δουλειά που γίνεται τελικά είναι χάσιμο χρόνο και αν θα φέρει καρπού. Είδαμε όμω ότι τα καταφέραμε και μπορεί να εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα στο Έσεξ, τα νοτιοανατολικά τη Αγγλία, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να επεκταθεί η ζωονόφο. Και γι' αυτό, νομίζω, και γι' νομίζω ότι θα πρέπει να ε, αγωνιστούμε όλοι στην προσπάθεια αυτή. Ο κύριο Μποβέ βλέπω να κουνάει το κεφάλι του και ξέρω ότι το πράσινο κίνημα δεν είναι υπέρ των εμβολιασμών, όμω σα διαβεβαιώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ζωτική σημασία να γίνουν εμβολιασμοί. Καλώ λέει ο Πρόεδρο. Και πριν δώσω το λόγο στον, κύριο στον Αντιπρόεδρο κ. Βαζερόφσκι, θα ήθελα να παρακαλέσω από την Επιτροπή τον κύριο Λαντόνα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όπως επίσης και όλους όσους πήραν το λόγο γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ομοφωνία από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξη των τεχνικών προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει επίσης συμφωνία και στο ότι υπάρχει ανάγκη να υιοθετήσουμε το κείμενο αυτό επιγόντω για να επιτρέψουμε να εκκινήσει ο εμβολιασμό πριν από το θέρο. Υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα προ επίλυση. Υπάρχει το θέμα των πινάκων αντιστοίχηση, σαν παράδειγμα εμείς έχουμε συμπεριλάβει το θέμα στην πρότασή μας και από δική μου πλευράς ελπίζω να υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γύρω από τους πίνακες αντιστοίχησης. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και υποστήριξαν τις θέσεις μου. Δεν μπορώ παρά να σας διαβεβαιώσω ότι ο κύριος γενικό μας στόχος είναι να προχωρήσουμε το χύτερο δυνατό σε αυτήν την έγκριση αυτής της οδηγίας, έτσι ώστε να δεθεί σε εφαρμογή εγκαίρω και να προχωρήσουμε στου εμβολιασμού. Από την άλλη βέβαια θα προσπαθήσω και να ε, υποστηρίξω και να επιδιώξω το άλλο, την άλλη επιδίωξη του ε, πίνακα αντιστοιχείων μέσα στον Απρίλιο ελπίζω να τα καταφέρουμε σε συνομιλίες με το Συμβούλιο, να πείσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα ως προς τους πίνακες αντιστοιχίας και στη τελευταία ανάλυση να προχωρήσουμε κατά τρόπο συνεπή με το προηγούμενο το οποίο έχουμε χαράξει, ε, ώστε να μπορεί και, η να είναι δυνατόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα νομοθετήματα να επισυνάπτονται αυτοί οι πίνακες αντιστοιχία ε, που δείχνουν πώς ακριβώς εφαρμόζεται μια οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Δεν πρέπει να είναι κάτι δύσκολο αυτό. Υπάρχουν πολύ πιο περίπλοκα νομοθετήματα, νομοθετήματα στο, στα οποία ήταν ίσω πιο δύσκολο να ενταχθεί ένα τέτοιο πίνακα αντιστοιχεία. Στην υπερσυγκεκριμένη περίπτωση όμω δεν βλέπω καμιά δυσκολία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε του στόχου μα. Κατά κύριο λόγο έχουμε να κάνουμε με το περιεχόμενο, δηλαδή τη δυνατότητα να προχωρήσουμε γρήγορα στην αξιοποίηση των εμβολίων. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μέχρι τις, ε, στις 7 Απριλίου μάλλον να υιοθετήσουμε την έκθεση για να προχωρήσει σε έγκριση. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της μισθές διατάξεως ε, για σήμερα το απόγευμα. Ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Εξέταση της προτάσεως ψηφίσματος προφορική ερώτηση για την αθλητικότητα των αντιβιωτικών έχει ως στόχο να επεκτείνει κάποια συστήματα επιτήρησης που ισχύουν σήμερα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας στον τομέα της κτηνοτροφίας. Η χρήση αυτών των αντιβιωτικών στα ζώα δεν ε, εποπτεύεται ικανοποιητικά. Εδώ ως ε, στο ψήφισμα, για το ψήφισμα μάλλον ως βάση χρησιμοποιείται το έγγραφο P7 τα 2010 130. Θα πρέπει λοιπόν το συντομό δυνατό να έχουμε ένα ψήφισμα σχετικά με την αυθεντικότητα στα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στα ζώα. Πρόκειται για μια εργασία την οποία θα κάνουμε ως Επιτροπή Γεωργίας, αλλά τι θα την προσυπογράψω εγώ, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Πόλσεν που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. Κύριε Αντιπρόεδρο Πόλσεν, να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη. Τα πράγματα προχώρησαν πολύ γρήγορα και ένα ψήφισμα που είχαμε δει στην Επιτροπή μας ε, το είδαμε στην Πράσινη Εβδομάδα. Μετά δεν μένανε παρά δύο μέρες για τη μετάφραση. Και έτσι το κείμενο δεν είναι πλήρες πρέπει να πω. Τα δεδομένα τα επιστημονικά δεν έχουν αλλάξει. Είχα μια συνάντηση στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα με τους κοιόδης ηγητές. Χρήσιμη, πολύ χρήσιμη. Πολλές ε, προτάσεις ε, τροποποίησης ακούστηκαν τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη στην πρόταση ψηφίσματος. Προτάσεις που αφορούν κυρίως τη δυνατότητα χρήσης των αντιβιωτικών. Και βέβαια ε, για τον άνθρωπο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό αφορά τους, ε, τα ζώα, την κτηνοτροφία. Στη σύγχρονη κοινωνία, στην Ευρώπη σήμερα, θεωρώ αδιανόητο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το ζώο να μην χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά τα οποία φέρουν αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν. Θέλουμε να διατηρήσουμε την δυνατότητα της χρήσης των αντιβιωτικών. Δεν πράξαμε όμως ένα σφάλμα. Ότι διαγράψαμε αυτή την ουτοπική ε, γνωμοδότηση ή τοποθέτηση μάλλον ότι δεν χρειάζονται τα αντιβιωτικά και ότι επιδιώκουμε το μέλλον της Ευρώπης να είναι απαλλαγμένο από αντιβιωτικά. Γιατί είναι τοπικό φυσικά κάτι τέτοιο. Εμείς όχι, αντιθέτως διαγράφουμε αυτή τη ε, διατύπωση. Ε, βλέπουμε το μέλλον της Ευρώπης όσο δυνατόν βέβαια χωρίς τη χρήση αντιβιωτικών, δηλαδή αναζητούμε τις εναλλακτικέ που θεωρούμε ότι θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε και την σημασία του να γίνονται έλεγχοι Η απαγόρευση δηλαδή χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία ή στην ανάπτυξη των ζώων, ε, δεν μπορεί να αφορά την ανάπτυξη των ζώων και αντιβιωτικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Εδώ είναι που δεν έχουμε τη γενική επισκόπηση, εδώ είναι που δεν έχουμε μια γενική ε, αντιμετώπιση, μια ε, ομοιόμορφη στάση στην χρήση των αντιβιωτικών. Ε, από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλες προτάσεις Διάφορες ομάδες έχουν διαφορετικές απόψεις. Η πράσινη Φερρυπίνη. Θα ήθελαν να ε, χρησιμοποιήσουν τον όρο βιομηχανική γεωργία ως ε, λόγο χρήσης ή ως κριτήριο χρήσης των αντιβιωτικών. Ενώ Άλλοι ζητούν ε, κριτήρια που να είναι για τους πάντες κοινά ε, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε όρους ευαίσθητους, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μια, με ένα κοινό ψήφισμα της Επιτροπής Γεωργίας, έτσι, δεν είναι δική μου η πρόταση, δεν είναι προσωπική έκθεση, πρόκειται για ένα ψήφισμα της Επιτροπής Γεωργίας, ένα ψήφισμα δηλαδή στο οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ή δυνατόν την ομοφωνία. Προσπαθώ λοιπόν να εξασφαλίσω συμβασμούς λέγοντας ότι οι μορφές κτηνοτροφίας, το είδος της κτηνοτροφίας που χρησιμοποιείται μπορεί να οδηγήσει σε μια ε, μεγαλύτερη συγκέντρωση και ως εκ τούτου κίνδυνο ε, επιμόλυνσης. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, στο κτίριο που βρισκόμαστε, με το air condition και ένα κοινό σύστημα air condition που ισχύει για ολόκληρο το κτίριο, προφανώ μπορεί να μεταδοθεί μειονόσο από τον ένα στον άλλον και ο ένα να μολύνει τον άλλον. Ε, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι έτσι οι συνθήκε τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια τα Προβλήματα παραμένουν, δεν είναι τόσο σημαντικά. Ευχαριστώ, Γκαρθία Μενές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σηκώνω την πρόκληση της κυρίας Πόλσεν και περιμένω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να αναζητήσουμε να βρούμε κάποια κοινά στοιχεία ως Επιτροπή. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει πάντως να εξορροπηθεί η πρόταση ψηφίσματος. Νομίζω πως το θέμα της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά θα πρέπει να εξεταστεί ομού με τα υγείας του ανθρώπου και της υγείας των ζώων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη στο ψήφισμα που εξετάζουμε, να γίνουν επίσης κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, έχουν να καταλήξουν. Στο σημείο 12 γίνεται αναφορά στις ε, μεταφορές ζώων και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται εδώ αναφορά στις μεταφορές των ζώων. Μεταφορές γιατί όχι εμπόριο σε και αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη, άλλη φάση και στάδιο της αλυσίδας. Έχουμε εδώ τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο ζήτημα, αλλά δεν ε, περιέχουν ε, πουθενά το ζήτημα της μεταφοράς των ζώων. Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να το συμπεριλάβουμε στο ψήφισμά μας. Όπως σας είπα, ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι ποικίλε απόψεις. Ευχαριστώ τα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν διότι έδειξε ιδιαίτερη προθυμία κατά την κατάθεση του ψηφίσματος. Είχα μια συνεδρίαση σχεδόν εισηγητών την περασμένη εβδομάδα και όντως είχε την ε, προθυμία, τη βούληση να καταγράψει και να δεχθεί τις θέσεις ε, των συναδέλφων. Υπάρχει μια σχέση άμεση ε, ανάμεσα στη χρήση αντιβιωτικών για τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, εξάλλου και στην τελευταία πρόταση αναφέρεται. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάψουμε να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά στην κτηνοτροφία. Αλλά πρέπει επίσης να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρήση των αντιβιωτικών είναι πολύ διαφορετικός στην κτηνοτροφία. Χρειάζεται λοιπόν να τονίσουμε πως ε, όταν θα έχουμε λάβει τα απαραίτητα στοιχεία από τα κράτη-μέλη πρέπει να τα εξετάσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να δράσουμε σε ενωσιακό επίπεδο, ίσως ε, με νέους κανόνες, ε, νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την απαγόρευση πώλησης κάποιων αντιβιωτικών και θα πρέπει να σκεφτούμε μια ενωσιακή λύση του προβλήματος. Τώρα, στις ε, μεταφορές ε, συμφωνώ. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε όλες τις ε, πτυχές που έχουν συνέπειες στην μεταφορά των βακτηρίων και των ιών, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και οι μεταφορές αποτελούν ένα κίνδυνο και τονίζω για μια ακόμα φορά ότι η συζήτηση ήταν πολύ ανοιχτή και σίγουρα θα καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η ε, κυρία Μαγκίνες. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Πόλση γιατί ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο σας έχει απασχολήσει πολλές φορές στην Επιτροπή. Είναι ισορροπημένε και βάσιμες ε, οι παρατηρήσει σας. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, να αντιληφθούμε τι συμβαίνει και να μειώσουμε στο βαθμό που είναι αυτό δυνατό τη χρήση των ε, εμβολίων. Κάποιες ε, παρατηρήσει στην τέταρτη παράγραφο, εκεί όπου λέει στο τελευταίο κομμάτι που γραμμίζει τη σημασία της εισαγωγής καλών στιμάτων καλών συστημάτων στην κτηνοτροφία. Η λέξη καλών με ενοχλεί, διότι υπονοεί ότι τώρα έχουμε κακά συστήματα. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε καλύτερα συστήματα παραγωγής κτηνοτροφίας κτλ. με μείωση δυνατών των ε, τη χρήση των εμβολίων. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό των μεταφορών. Άρθρο 12 λοιπόν, όπου πάλι η διατύπωση αναφέρεται σε, αν, σε ανεκτές συνθήκες ή αποδεκτές ε, μεταφοράς. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ εύστοχη διατύπωση, διότι ε, αν εφαρμόζουμε τους κανόνες περί μεταφοράς των ζώων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συνεπάγεται και ε, κατάρτιση του προσωπικού ανά την Ευρώπη στην διαχείριση του άγχους των ζώων, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με την ευημερία και την υγεία αυτών. Παράφωση παριθμών 7 προβλήματα με την ΕΦΑΟ και την ΕΦΣΑ, ζητήματα που ενδεχομένω να προκύψουν και που ίσω να έχουν και δημοσιονομικέ επιπτώσει, πρέπει να τα δούμε. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε συμβαστικέ ε, λύσει, σε συνεργασία όλοι του κοιόδη. Σα θυμίζω εδώ ότι οι τροπολογίε θα πρέπει να κατατεθούν. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η Ελίζα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την στράτευσή σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα στη συνάδελφο για τις προτάσεις της. Όντω το κομμάτι το σχετικό με τις μεταφορές ε, των ζώων και των συστημάτων ε, κτηνοτροφίας είναι, αυτό το, στο οποίο αυτά στα οποία χρειάζεται μια καλύτερη διατύπωση. Ταυτόχρονα ωστόσο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια κατάσταση, φερειπίν στις μεταφορές ε, ζώων, όπου πέραν της, του μελήματος για την εφημερία των ζώων μπορούμε με μια καλύτερη αντιμετώπιση της μεταφοράς να εμποδίσουμε τη διάδοση ζωονόσων. Ε, Άρα έχουμε και αυτό το όφελος. Βέβαια το ζήτημα είναι το πώς θα διατυπώσουμε το κείμενο έτσι ώστε να είναι αποδεικτό για όλους. Και θα ήθελα να πω ότι... Ε, η πρόταση περί συλλογής καλύτερων δεδομένων ή ανάλυση τους ε, ή παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιωτικών ως υπέρτατου στόχου και ε, της αξιοποίησης των ε, αντιβιωτικών ως, ως αποτελεσματικού μέσου για την αντιμετώπιση των ζώων νόσων και των νόσων, νομίζω ότι ε, ίσως χρειάζονται μια κάποια ένα κάποιο χτένισμα όπως είπε, ένα λουστράρισμα, αλλά πάντως εξασφαλίζουν μια, ε, ένα κείμενο ψηφίσματος πολύ καλό. Και μπορεί να έχουμε συζητήσει ε, θέματα ε, απαγόρευσης των αντιβιωτικών στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές καλύτερα, ε, και εν τέλει να οδηγηθήκαμε στον μεγάλο προβληματισμό σχετικά με την ε, ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ε, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα καλό ψήφισμα και ευχαριστώ πολύ την ε, συνάδελφο για τη συνεργασία. Ευχαριστώ, Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν για την εξαιρετική δουλειά της και για τη συνάντηση που οργάνωσε στο Στρασβούργο. Εγώ δεν ήμουν παρόν, αλλά ένας από τους συνεργάτες μου πήγε. Θα ήθελα ε, για δύο θέματα να κάνω μία παρατήρηση γιατί δεν ε, ίσως ε, παρουσιάζονται σωστά στο έγγραφο. Επιστημονικά γνωρίζουμε σήμερα ότι η συγκέντρωση ζώων σε μεγάλα κέντρα οδηγεί στην αύξηση της χρήσης των αντιβιωτικών. Αυτά είναι επιστημονικά στοιχεία τα οποία μας δίδουν τα Υπουργεία των χωρών μας. Είναι μια πραγματικότητα που έχει σχέση με το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Το επόμενο θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε μια θέση σαν Ευρωπαίοι είναι το θέμα της υγείας των γεωργών και των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτά τα ατελειέ ουσιαστικά λέει ο μιλητής αυτοί παρουσιάζουν σήμερα τη μεγαλύτερη αντίσταση στα αντιβιωτικά γιατί σπνέουν κόνη τροφίμων και το γνωρίζουμε από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από, από το Ταμείο πρόνοιας των γεωργών στη Γαλλία ότι παρουσιάζουν τεράστια αντίσταση στα αντιβιωτικά γιατί αναπνέουν τις ουσίες αυτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα παρατηρητήριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε το σύνολο της μελέτης αυτής να το αντιμετωπίσουμε γιατί πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας και δεν θα είναι σε θέση να θεραπευτούν. Πρέπει λοιπόν αναχώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίσει το τι βιώνουν οι γεωργοί σχετικά με την αντίσταση στα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή ζώων. Ευχαριστώ Ζωζέ. Άγνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανησυχώ λίγο για υπερβολική νομοθεσία στον τομέα αυτό, για όλους εμάς που παράγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα, συμμετέχουμε σε ασφαλιστικά προγράμματα που μας απαγορεύουν να χρησιμοποιούμε χωρίς έλεγχο αντιβιωτικά. Πρέπει να υπάρξει ε, συνταγή ε, κτηνιάτρου για την καταπολέμηση μιας ασθένειας η οποία έχει γίνει αντικείμενο δια... Ε, διάγνωσης. Και δεν θέλω οι πολιτικοί να ανακατεύονται στα πόδια μας. Σχετικά με τη μεταφορά. Και εδώ ανησυχώ για την έτσι, υπερβολικά αγαθή πρόθεση ορισμένων. Στην Αγγλία έχουμε μια στρωματοποίηση της βιομηχανίας που ασχολείται με, το πρόβιο κρέας. Δεν θέλουμε εμείς να υπάρξει υπερβολική νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε έτσι και αλλιώς και χώρους απομόνωσης για τα ύποπτα ζώα. Παρακαλώ λειτουργεί το σύστημα, μην μας ανακατεύετε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, τον κύριο Βαντάικ. Και μετά θα κλείσει η κυρία Πόλσον και θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον δήμαρχο Φερντινάντο Αλμπάνο, δήμαρχο της πόλης Μπρατσιλιάνο, της ορεινής περιοχής αυτής που παράγει κεράσια. Τους α, χαιρετίζω λοιπόν. Ο κ. Βαντάκη έχει το λόγο. <clears throat> Good afternoon. Yes, I just want to very briefly. Ευχαριστώ. Ε, πολύ σύντομα. Θα ε, να ευχαριστήσω. Είναι ένα θέμα περίπλοκο και εμεί από την Επιτροπή προσπαθούμε να ε, διατυπώσουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Όπω είπαν και πολλοί από του ομιλητέ εδώ, δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένες δράσεις ε, το πρόβλημα, το και ως εκ τούτου σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε μια ανακοίνωση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων με μακροπρόθεσμων με σημαντικά θέματα που έχουν ήδη υπογραμμιστεί, η Φερρυπίν συλλογή δεδομένων, ε, μια βάση δεδομένων που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για να δώσει και καθοδήγηση στην ε, πολιτική μας, αλλά ταυτόχρονα και επιτήρηση που υπογραμμίζει ιδιαίτερος το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, περιμένω λοιπόν να δω το τελικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Βαν Ντάικ. Η αντιπρόεδρος κυρία Πόλσον έχει το λόγο. Και επειδή τελειώνουμε έγκαιρα, θα ήθελα να συνεδριάσουμε αυτής αμέσως ε, μετά με τους συντονιστές και άλλα αύριο θα ξεκινήσουμε 9.45. Κυρία Πόλσε. Ευχαριστώ και τον Ζε Μποβέ, ε, διότι εξήγησε πως ε, Εάν όσοι εργάζονται στον τομέα της γεωργίας πέσουν θύματα των βακτηρίων των ανθεκτικών και το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς μετά είμαστε τα σήματα διότι ούτως έχει τροφική αλυσίδα. Διότι με την εμπορία, με την μεταφορά νέων ζώων, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να παίρνουμε 10, 15, 20 παιδιά και να τα βάλουμε στην ε, ίδια τάξη. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, τάξεις ε, με παιδιά εάν δεν έχουμε στη διάθεσή μας αντιβιωτικά. Διότι είναι αυτά τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τους ποικίλου ιούς. Αυτό είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται να το λάβουμε υπόψη. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς ζούμε τις επιπτώσεις της φύσης. Η παραγωγή χείρων δεν έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στα νοσοκομεία από τις ε, κεντρικές πόλεις, σύρες, διότι είναι φορείς μικροβίων τα οποία δεν καταπολεμούνται εύκολα. Όπως όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Χρειάζομαι λοιπόν να είμαστε σαφείς για να εξηγήσουμε πως η ε, κατάσταση είναι γνωστή φυσικά σε όλους, αλλά ουδής ασχολείται με την ουσία του προβλήματος. Αυτά είναι η κατάσταση λοιπόν χρειάζεται να αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Τέρμα στα ωραία λόγια, αυτό που χρειάζεται είναι δράση. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Πόλσεν. Νομίζω πως υπάρχει ευρύτατη σύγκληση θέσεων και απόψεων. Να σας υπενθυμίσω πως αύριο η συνεδρίαση της Επιτροπής μας προβλέπεται στις 9.45, όπως προείπα. Θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με τις ψηφοφορίες και μην ξεχάσετε να φέρετε τις κάρτες σας γιατί θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 5 λεπτά διακοπή και μετά συνεχίζουμε με τους συντονιστές. Μα μουλιούς μα σε τα μου τι; <laughs>